Bonjour à toutes et à tous. Καλή σα ημέρα. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης και ε, με τα χαράς υποδέχομαι τον πρόεδρο της Έχνωσης Λέψεως, κύριο Σόρος. Περνάμε στην έκθεση με τις διατάξεις mm. και την έκθεση αυτής Υπάρχει μια αλλαγή στην μέσα διάταξη. Ο κ. Νόησερ θα μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του σχετικά με το πρωτόκολλο αλίας με το κύριο Μπάτι σήμερα. Και αν για αύριο προέρχεται μια τροποποίηση επίση τη μεσαία διατάξεω και η σειρά των σημείων θα είναι εξή. Θα ξεκινήσουμε από την νομοδότηση κυρία Κρετού, ε, φιλοκτονία των ε, γυναικών θα συνεχίσουμε με την έκθεση Κάσμαν για την υγεία και τα δικαιώματα αναπαραγωγής. Μετά περάσουμε την έκθεση Καμίνσκι, ε, διαφθορά στον δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό συνέπειε στα δικαιώματα των ανθρώπων στις τρίτες χώρες. Μετά έκθεση ΡΟΑΤΑ για την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην περιοχή της, Κουσαέλ. Και θα ολοκληρώσουμε τις πρωινές εργασίες με την νομοδότηση του κυρίου Κάσμαρέκ για την ποιότητα των καυσίμων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν σχόλια επί της μισής Εφόσον δεν υπάρχουν, τότε εγκρίνεται όπως έχει τροποποιηθεί. Έχετε λάβει τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 23 Απριλίου 2013. Αν έχετε παρατηρήσεις αναφορικά με τα εν λόγω πρακτικά, παρακαλώ να τα ενημερώσετε τη γραμματεία πριν από το τέλος της συνεδριάσεώς μας. Ιδάλλως τα πρακτικά θα εγκριθούν ως έχουν. Λάβατε επίσης σωστές τις και τις αποφάσεις που λάβαμε κατά τη διάρκεια των συντονιστών στις 22 Απριλίου 2013. Αν έχετε παρατηρήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα αυτής της συνεδρίασης, παρακαλώ ενημερώστε την γραμματεία πριν από την ε, λήξη της συνεδριάσεως. Ιδάλλως ε, τα πρακτικά, τα αποτελέσματα μάλλον θα εγκληθούν όσοι έχουν. Δύο ανακοινώσεις έχω να σας κάνω. Η πρώτη αφορά της ε, ψηφιακής υπογραφής και τον ρόλο της Κομισιόν μας ως, ως Επιτροπής Πιλότου στο ζήτημα. Η Επιτροπή μας καταβάλει προσπάθεια μαζί με τις χώρες που με τις ε, επιτροπές που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική ε, υπογραφή προκειμένου να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανή διαδικασία. Εν τω μεταξύ θα έχουμε το χρόνο, την δυνατότητα μάλλον από την επόμενη εβδομάδα να υπογράφουμε ή να συνυπογράφουμε ε, ε, ε τροπολογίες στις εκθέσεις και νομοδοτήσεις μας. Και δεν θα χρειάζεται να στέλνονται μέσω τηλεμιοτυπίας. Βρείτε ε, τις πληροφορίες στο e-committee, αλλά θα λάβετε και μια πληροφόρηση για μια ενημερωτική συνεδρίαση που θα οργανωθεί στις 6 Ιουνίου. Να σας ενημερώσω επίσης ότι έλαβα σήμερα, μάλλον συνάντησα σήμερα μια αντιπροσωπεία του ΟΗΕ των προσφύγων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Συρία. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η κατάσταση είναι τραγική και επέσταν την προσοχή της Επιτροπής μας για την ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί. Υπάρχει μια τεράστια ροή προσφύγων και υπολογίζονται σε 3,5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες εκτός Συρίας μέχρι τα τέλους του έτους. Ένα εκατομμύριο στην Ιορδανία, ένα εκατομμύριο στο Λίβανο, στην Τουρκία επίσης, αλλά και μια εκατοστή χιλιάδες πρόσφυγες στο Βόρειο Ιράκ. Υπάρχουν πάνω από 4 εκατομμύρια πρόσωπα στο ιστορικό της Συρίας που εξαρτώνται από την διανομή τροφίμων έχουν ανάγκη από 16 εκατομμύρια ανά εβδομάδα μόνο και μόνο για να τραφεί ο πληθυσμός αυτός. Τα χρήματα λείπουν και κάνουν έκκληση σε εμά, αλλά γνωρίζουμε τους περιορισμούς για τις περικοπές στον προϋπολογισμό μας. Κάνω έκκληση λοιπόν προς εσάς βουλευτές, ώστε στις χώρες σας να αναλάβετε τα απαραίτητα διαβήματα, ώστε να λάβονται περισσότερα χρήματα για την ζωτική σημασία δράση του οργανισμού που σώζει ζωές στην Συρία. Η Κομισιόν έχει κάποια ανακοίνωση να μας κάνει. Ναι. Ο κύριος Πίτερ Κρέγκ Μακουάιρ έχει το λόγο από την Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία. Καταρχήν η Κομισιόν ενέκρινε μια ανακοίνωση στις 15 Μαΐου για τις τοπικές αρχές. Ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι ενισχύοντας τις τοπικές αρχές για την προαγωγή της διακυβέρνησης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές παίζουν ρόλο κλειδί στην χρηστή διακυβέρνηση και την υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο και προκειμένου να ανακοθεί το πλήρες δυναμικό αυτών των περιοχών θα πρέπει να εστιάσουν, εστιάσουμε στην λήψη αποφάσεων για θέματα ανάπτυξης. Τώρα προχωράμε με τις εργασίες σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης από το Συμβούλιο. Δεύτερον, η Κομισιόν ενέκρινε μια ανακοίνωση στις 21η Μαΐου για την θανάστευση που φέρεται τον τίτλο μεγιστοποιώντας ε, τις επιπτώσει ε, ε, της μετανάστευσης και αυτό αποτελεί τη βάση για μια κοινή θέση της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγγνώμη, στον διάλογο που διεξαχθεί στον φθινόμπορο στον ΟΗΕ για το ζήτημα της μετανάστευσης είναι κάπως επίγον ζήτημα και θα πρέπει να υπάρξει μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά στόχος είναι να προάγουμε την κινητικότητα της μετανάστευσης ως ε, και την ε, πρόθεσή της προς τις ε, επιθυμητές κατευθύνσεις. Επίσης, ως σε ό,τι φορά τη δέσμη για το 11ο πακέτο έχουμε προτείνει ένα νέο πρωτόκολλο για τη συμφωνία με το Κοτονού και αυτό θα περάσει από το Συμβούλιο του Υπουργού Εξωτερικών αύριο. Αυτές ήταν οι τρεις ανακοινώσεις που θα σας κάνω. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Δεν έχουμε λάβει ερωτήσεις προς την Κομισιόν κάτι το οποίο μας επιτρέπει να περάσουμε στο έβδομο σημείο της Μερσίας Διατάξεως, δηλαδή ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Κίκ Κικμπαφόρη Σόρο, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Ακτής του Ελεφαντιστού, που είχα την χαρά να τον συναντήσω ήδη και θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τις προοπτικές στην ακτή του Ελεφαντοστού. Όπως γνωρίζετε, αυτή του ελεφαντοσού έχει κάποια πρόοδο μετά από την μετεκλογική κλίση του 2010-2011, ακόμα και αν μεγάλες προκλήσεις παραμένουν. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής θα ήθελα, Πρόεδρε, να σας ενθαρρύνω στο να συνεχίσετε τον πολιτικό διάλογο, ο οποίο περνάει ε, αναμφιβόλως και από το σώμα του οποίου προεδρεύεται. Δεν θα τονίσουμε αρκετά τον ρόλο της Εθνικής Εθνικής στην δημοκρατία. Σας παροτρύνουμε λοιπόν να θέσετε στη μέση διάταξη των συζητήσεων τα μεγάλα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην βάση της κρίσης που έπληξε τη χώρα σας, ειδικά το ζήτημα της ισορροπίας των εξουσιών, την δυνατότητα ανάπτυξη του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον διάλογο για την συμφιλίωση και τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί σε αυτές τις εργασίες ή ακόμα και στο ζήτημα των, ε, της διανομής της γης. Αυτά είναι, λοιπόν είναι κάποια ζητήματα πρώτα τα οποία θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας ε, σήμερα. Έχετε το λόγο για 20 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να αρχίσω πρώτα απ' όλα με ευχαριστίες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε η αντιπροσωπεία δηλαδή της ακτής ελεφαντοστού εκ μέρους του λαού της χώρας που μας δίνεται τη δυνατότητα να έρθουμε και να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Είμαι επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας βουλευτών από πέντε κοινοβουλευτικές ομάδες από την ακτή Ελεφαντοστού. Στην Εθνική Συνέλευση εδρεύουν 255 βουλευτές. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρέσβη της Αυστρίας και τον πρέσβη της ακτής Ελεφαντοστού που βρίσκονται εδώ στις Βρυξέλλες. Όπως καταλαβαίνετε τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον λόγο των αντιπροσώπων των λαών όταν αυτοί μιλούν για το μέλλον τους. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ εμένα και την Εθνική Συνέλευση της Ακτής Ελεφαντοστού να έρθουμε εδώ και να πάρουμε το λόγο μπροστά σας. Και παίρνω το λόγο σήμερα μπροστά σας, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, είναι γιατί η κρίση στη χώρα μου έληξε. Σήμερα οικοδομούμε το κράτος δικαίου, οικοδομούμε τη δημοκρατία στην ακτή ελεφαντοστού. Όπως είπατε κι εσείς, είναι αλήθεια ότι παραμένουν πολλές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές, πρέπει να σας πω, είναι ακριβώς εκείνες που έχει κάθε χώρα που βρίσκεται στη διαδικασία της ανάπτυξης. Κάθε χώρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες προκειμένου να παλύψει την ένδια. Είναι χαρακτηριστικό κάθε χώρα σε οποία προσπαθεί να βγει από μια κατάσταση ένδιας η οποία ίσχυσε για δεκάδες χρόνια όπως έγινε στη χώρα μου. Πολιτικά μιλώντας τώρα, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι η ακτή λειτουργεί κανονικά. Όλοι οι θεσμοί της δημοκρατίας έχουν καθιδρυθεί. Μετά την μετεκλογική κρίση, τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί. Έξι μήνες μετά, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τη μεγάλη κρίση, καταφέραμε να οργανώσουμε κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες κατέληξαν στην ε, καθίδρυση της Εθνικής Συνέλευσης της Ακτής του Ολεφαντοστού, όπως σας το περιέγραψα πριν. Στη συνέχεια, συνεχίσαμε και επιμείναμε στις προσπάθειές μας προκειμένου να οργανώσουμε δημοκρατικές τοπικές εκλογές που να διέπονται από διαφάνεια. Δημοτικές πρώτα απ' όλα και περιφερειακές στη συνέχεια, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μέσα σε ένα ειρηνικό κλίμα. Και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν μια πρόκληση που αντιμετώπιζε τόσο η κυβέρνηση όσο και ο της χώρας. Οι τελευταίες λοιπόν τοπικές εκλογές συμπληρώνουν, ολοκληρώνουν τη μακρά εκλογική διαδικασία και με μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να σας πω σήμερα πως τα πράγματα πήγαν καλά. Βέβαια, κυρία Πρόεδρε, μπορούμε να καταδικάσουμε το γεγονός ότι δεν συμμετείχαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Το ΕΣΠΗ, για παράδειγμα, που είναι το κόμμα του προηγούμενου πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στα χέρια της διεθνούς δικαιοσύνης. Ο λόγος, ο οποίος αναφέρθηκε, είναι ότι πρώτα έπρεπε να ελευθερώσει τον τέος πρόεδρο η διεθνής δικαιοσύνη και μετά να μπουν στην πολιτική διαδικασία και να συμμετάσχουν στις εκλογές. Κάτι το οποίο θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι δεν είναι κάτι που εξαρτάται από τις αρχές της χώρας, γιατί ο κύριος Μπάκμπο είναι στα χέρια της διεθνούς δικαιοσύνης. Για μας τώρα, που είμαστε Εθνική Συνέλευση της Ακτής Ελεφαντοστού, η πολιτική της άδεια καρέκλας δεν είναι κάτι καλό. Και οι κυβερνώντες, ε, τα κόμματα της πλειοψηφίας, της μειοψηφίας έχουν το δικαίωμα να προχωράνε σε μια πολιτική που να τους συμπεριλαμβάνει όλους, αλλά άλλο τόσο και η, μειοψηφία πρέπει να συμμετέχει στη δημοκρατική διαδικασία. Από πλευράς ασφάλειας τώρα, πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Μετά την μετεκλογική κρίση, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου είχαν αποδυναμωθεί κάπως και έτσι Σήμερα βελτιώνουμε και έχουμε την αστυνομία και την χωροφυλακή, την εθνική χωροφυλακή που είναι πραγματικά πρώτης τάξης. Ο στρατός επίσης αναδιαρθρώνεται. Τώρα για να εκτιμήσουμε καλύτερα πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση ασφάλειας στη χώρα, σας λέω ότι ο γενικός δείκτης ανασφάλειας έχει περάσει από το επίπεδο στο επίπεδο του 1,6. Κάτι που σημαίνει ότι οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να επιστρέψουν, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης, που σήμερα περιμένουμε στην ακτή Ελεφαντοστού. Για μια χώρα σαν τη δικιά μου, που έχει γεωστρατηγική σημασία θέση στην Αφρική, η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλη. Γιατί στα σύνορά μας βρίσκεται το Μαλί. Και ξέρετε τι προβλήματα υπάρχουν ε, ασφάλεια στο Μαλί. Δυτικά έχουμε τη Λιβερία. Και ξέρετε ότι η Λιβερία είναι μια χώρα που και εκείνη βρίσκεται σε κατάσταση αστάθειας. Οπότε το θέμα της ασφάλειας αποτελεί προτεραιότητα για την ακτή ελεφαντοστού. Και γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε, εμείς πιστεύουμε ότι η διεθνής κοινότητα συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε για το θέμα της ασφάλειας όχι μόνο στην ακτή του αλλά σε ολόκληρη την περιοχή. Ακριβώς επειδή υπάρχουν μεγάλες απειλές που δεν είναι οι συνήθεις απειλές που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα, είναι πολύ πιο ισχυρές, όπως είναι η τρομοκρατία στο Μαλί, για παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι θα έπρεπε να το προσέξετε αυτό το θέμα και εσείς όλους ιδιαίτερος. Οικονομικά τώρα. Η ακτή φαντοστού έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Είμαστε σε στάδιο οικονομικής ανάκαμψης στη χώρα. Πολλοί επενδυτές μετά τις μεταρρυθμίσεις, τις οικονομικές που κάναμε, ιδιαίτερα το πρόγραμμα που είχαμε μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές ε, Νομισματικό Ταμείο, καταφέραμε να φτάσουμε στο σημείο όπου η ακτή να είναι μια χώρα η οποία να καλύπτει τον επενδυτικό κόσμο και για το 2012. Και εδώ κοιτάξτε τα επίσημα στοιχεία τα οποία δίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ίδιο που λέει ότι έχει 9,8% ε, του ΕΠ ανάπτυξη η χώρα μας. Για το 2013 έχουμε επίσης πρόγραμμα και ξέρουμε ότι θα είμαστε στο 9% όσον αφορά την ανάπτυξη. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ένδια γιατί ξέρετε ότι κυρίως αγροτική χώρα είμαστε. Είμαστε η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής κακάο. Έχουμε τεράστιες καλλιέργειες, όπως επίσης νουακ καζού. το φιστίκι κάσους. Έπειτα, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια χώρα που έχει περάσει από πόλεμο, καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς γίνονται κάποια στραβοτιμονιές μερικές φορές. Όμως, ο πρόεδρος Κατάρα προσπαθεί να σταματήσει το φαύλο κύκλο της ατιμορρησίας που κυριαρχούσε στη χώρα για δεκαετίες και αποφάσισε να δημιουργήσει μια επιτροπή ερευνητική η οποία θα ρίξει φως σε όλα τα εγκλήματα τα οποία έλαβαν χώρα μετά την μετακλογική κρίση. Η επιτροπή αυτή λειτουργήσε και έδωσε την έκθεσή της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την έκθεση αυτή την έστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι εκείνο το οποίο θα δώσει συνέχεια στην έκθεση αυτή. Η Εθνική Συνέλευση, όσον αφορά εμάς τουλάχιστον, Εμείς από το 2011 είμαστε... Έχουμε τα ενία της χώρας φροντίζουμε για τους νέους νόμους και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην εθνική συμφιλίωση. Όλοι είναι παιδιά της χώρας. Όταν μια χώρα βγαίνει από ένα τέτοιο τραύμα όπως αυτό που ζήσαμε εμείς, είναι πολύ σημαντικό για όλους τους θεσμούς και επιμένω για όλους τους θεσμούς και για την εθνική ασφάλεια ο καθένας να παίξει το ρόλο του για να υπάρξει αυτή η συμφιλίωση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς επιμένουμε στο διάλογο και στο έργο της Επιτροπής αυτής όπως έγινε και στην Νότια Αφρική. Είναι μια δουλειά βέβαια που παίρνει πολύ χρόνο. Η Εθνική Συνέλευση παίζει και αυτή το δικό της ρόλο. Πιστεύουμε πάντως πως υπάρχουν αποτελέσματα, γιατί μετά τις προεδρικές εκλογές μπορέσαμε να οργανώσουμε και άλλες εκλογές οι οποίες έλαβαν χώρα μέσα σε ένα κλίμα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα εντελώς διαφορετική από αυτή που είχαμε μέχρι τότε. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να μπω και σε πολλές λεπτομέρειες. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι να τονίσω το εξής. Σήμερα, εδώ στην Επιτροπή σας μπορώ να πω και να επιμείνω για το ότι η εκτή ελεφαντοστού έχει μπει στο σωστό δρόμο. Εμείς παίζουμε το ρόλο που μας πρέπει στην Αφρικανική Ήπειρο και ελπίζουμε ότι θα αναλάβουμε στην ε, Νοτιοδυτική Αφρική επίσης τον ρόλο μας. Ο πρόεδρός μας εξάλλου προεδρεύει και το ΣΕΝΤΕΟ που συμμετέχουν οι κοινότητες των χωρών της Νοτιοδυτικής Αφρικής. Όλα τα στοιχεία τα οποία σας ανέφερα εννοείται ότι είναι στη διάθεσή σας να μπείτε σε περισσότερες λεπτομέρειες εφόσον το επιθυμείτε. Είμαι στη διάθεσή σας λοιπόν για ό,τι ερωτήσεις έχετε να μου κάνετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> Οι κύριοι βουλευτές έχουν το λόγο. Ο κύριος Πόγκα πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Εθνοσυνέλευσης της Ακτής του Ελεφανταστού, ευχαριστώ για την τιμή μου κάνετε να είστε σήμερα ανάμεσά μας. Θα ήθελα να έχω κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία συμφιλίωσης που αναφέρατε ότι εξάγεται στην χώρα σας. Η Επιτροπή Διαλόγου για την Συμφιλίωση που συστήσατε τον Ιούλιο 2011 εργάζεται με τρόπο ουσιαστικό. Αυτό θα ήθελα να γνωρίζω. Η πρόοδος είναι ουσιαστική. Το αναφέρω αυτό διότι η έκθεση που δημοσίευσε η Amnesty International στις 26 Φεβρουαρίου ενεστώντος έτους αναφέρει ότι η συμφιλίωση είναι δύσκολη στο μέτρο που πολλές ε, παραβιάσεις ε, γίνονται και κατά του κ. Μπακμπό από, την, από το στράτευμα παραμένουν ατιμόρυτες. Πώς λοιπόν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια συμφιλίωσης και επίσης η ε, Εθνική Επιτροπή Έρευνα ε, ε, έβαλε μια έκθεση για την μετά, την, τον, μετά τις εκλογές περίοδο. Μπορείτε να μας πείτε τι συνέχεια δόθηκε σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μισελ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας... Μάλλον, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας συγχαρώ και μέσω ημών και τις αρχές της αρχής του Ελφαλωτίου που πράγματι έβαλαν πάλι σε τροχιά την χώρα. Δεν υπάρχει εμβολία ότι πολλά πράγματα μένουν ημιτελή. Είχατε την αντικειμενικότητα να το πείτε στους ίδιους. Ε, τώρα ε, η ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί στην ε, ευθύ του είναι τόσο σημαντική που μας δείχνει ότι είναι ένας ε, εταίρος ε, σίγουρος, σταθερός στην περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να το τονίσω. Δεύτερη ερώτηση. Αυτά που σας είπα πρόκειται για συγχαρητήρια και θα πρέπει να συνεχίσετε. Να σας θέσω τώρα όμως μια ερώτηση σχετικά με το 9 9,5% ανάπτυξη έχετε τα απαραίτητα μέσα ώστε θα μπορέσετε, να μπορέσετε να βοηθήσετε την εκπαίδευση, την κοινωνική κατάσταση αλλά και όλα τα άλλα ζητήματα που άπτονται τους ε, κοινωνίας. Σίγουρα έχετε κάποια προγράμματα αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε μερικά πράγματα παραπάνω από σας. Και γιατί την παρατήρηση θέλω να γνωρίζω γιατί το FPI ε, παίζει, χρησιμοποιεί μάλλον την ε, πολιτική της κενής έδρας. Ε, το έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν από άλλες, σε άλλες περιπτώσεις. Το να απαιτήσουμε λοιπόν την την παράδοση του κυρίου Μπαγμπό ξέρετε ότι δεν είναι και τόσο ορθό να συμβεί πριν από το τέλος της διαδικασίας. Τι κάνετε εσείς ως πλειοψηφία για να αποδεσμευθεί η κατάσταση και για να οδηγήσετε το πρώην κόμμα του κ. Μπαγμπό σε αυτή τη διαδικασία της συμφιλίωσης. Παρακολουθώ τις εξελίξεις ε, στην αυτή του σε αυτή του ευχαριστώ, αλλά βλέπω ότι πρόκειται και για μια στρατηγική μάλλον της αντιπολίτευσης που δεν επιθυμεί να τεθεί σε τον μηχανισμό αυτών της συμφιλίωσης. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πρέπει να ζήσουμε αυτό, αλλά η πλειοψηφία πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια για να προσελκύσει αυτόν τον ε, κόμμα σε έναν ενάρετο κύκλο για την περαιτέρω συμφιλίωση. Αυτά είχα να πω. Το ε, τρίτο στοιχείο. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω αναφορικά με τις δυσκολίες που συναντάτε για την επιχείρηση DDR. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση πολύ λεπτή, γνωρίζω τις δυσκολίες αυτής της επιχείρησης, ειδικά στην επίδοση Φαρεστού. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε για τον αφοπισμό ε, και την επανένταξη. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Ίσως να μας πείτε κάτι παραπάνω για τις κοινωνικές πτυχές, ε, την παιδεία κλπ. Εντάξει, καλό είναι να, μιλάμε, να δημιουργούμε πλούτο και ευημερία, αλλά ένα κομμάτι αυτή τη ευημερία θα πρέπει να πάει προ την βελτίωση της, ε, του βίου των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να χαιρετήσω εδώ μια ομάδα επισκεπτών. Είναι προσκεκλημένη του κ. Γκέρενς στα πλαίσια της φιλίας Λουξεμβούργου-Πορτογαλίας. Καλώς ήρθατε. Είσαστε εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν και μαθητές από το German School of Brussels. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Ο κύριος Κόρτες Γάστρα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Πρόεδρε Σόρο. Ναι, περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας. Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Σας έχουμε εδώ, μπορούμε και να σας ακούσουμε και ελπίζω και στο μέλλον να υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με την ακτή ελεφαντοστού. 500 εκατομμύρια νομίζω είναι το ποσό που δίνει. Τώρα, το ακούσαμε ότι το 2012 είχατε 9,8% ανάπτυξη και ότι θα συνεχιστεί. Ωραία. Για την ανάπτυξη αυτή όμως έχουμε την αίσθηση ότι δεν φτάνει στον κόσμο. Φαντάζομαι ότι και εσείς το βλέπετε αυτό. Πιο πολύ από ό,τι το βλέπουμε εμείς ένας στους τέσσερις κατοίκους ζει κάτω από το όριο της ένδυας. Συνεπώς, θέλω να ξέρω τι πολιτικές εφαρμόζετε εσείς για να καταπολεμήσετε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή την απάλληψη της ένδυας. Και κάτι άλλο που νομίζω ότι μπορούμε μαζί να κάνουμε πρέπει να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο υπέρ της συμφιλίωσης. Να μην υπάρχει ατιμερησία και να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους, ίδια δικαιοσύνη για όλους. Πάνω σε αυτό το δρόμο νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασια μεταξύ μας. Έπειτα πριν από μερικές μέρες η Διεθνής Αμνηστία διαπίστωσε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στις καταχρήσεις που έγιναν πριν από πολλά χρόνια από το στρατό και ότι υπάρχει ένα αθρεμπόριο όπλων. Θέλω λοιπόν να ξέρω τι πρωτοβουλίες παίρνετε εσείς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Κατά τα άλλα και πάλι σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η καλή κοινοβουλευτική σχέση ανάμεσα δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Ακτής Ελεφαντοστού. Πρόεδρε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές και μετά θα περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Από τις ερωτήσεις σας είμαι ευτυχής και περήφανος που βλέπω ότι σας ενδιαφέρει η χώρα μου. Και με εκπλήσει επίσης πόσα πολλά πράγματα γνωρίζετε για την κατάσταση στο εσωτερικό της ακτής Ελεφαντοστού. Τώρα για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα αναφερθήκατε στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που αναφέρει ε, διάφορα, διάφορες παραβιάσεις που έχουν γίνει και αναφέρει το θέμα της ατιμορρησίας στην ακτή ελεφαντοστού. Ε, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που έχουμε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας πρέπει να ξέρετε ότι έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία η ο πρόεδρος της χώρας και εγώ πρόεδρος του Κοινοβουλίου για ανθρώπους που λέω ότι είναι πολιτικοί πρόσφυγες η Διεθνής Αμνηστία, καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι από τους πρώτους που λέω ότι πρέπει να δώσουμε σημασία στην έκθεση αυτή, γιατί και εγώ από τη Διεθνή Το πραγματικό πρόβλημα δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα θέματα τα οποία αναφέρει η Διεθνή Αμνηστία. Σας λέω μάλιστα ότι μετά τις εκλογές η κρίση στη χώρα μου είχε σαν αποτέλεσμα πάνω από 3.000 νεκρούς σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η Προεδρία της χώρας μόνο το 2011 όμως μπόρεσε να ασχοληθεί. 1η Ιουνίου του 2011 ανέλαβε κυβέρνηση. Στο μεταξύ όμως τι έγινε, δεν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν υπήρχε δικαστήριο. Οι δικαστές διώκονταν, είχαν φύγει. Ο κόσμος ανακαζόταν να εγκαταλείψει τα σπίτια του. Χρειάστηκε να ξαναφτιάξουμε το κράτος και τους θεσμούς. Και σας το είπα, 1η Ιουνίου του 2011 δεν βρήκαμε θεσμούς, πέρα δηλαδή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που εκλέχτηκε. Τον Απρίλιο λοιπόν του 2012 ε, μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την εκλογική διαδικασία. Συνεπώς, αυτά που λέει η Διεθνής Αμνηστία, όλες οι παραβιάσεις και υπερβολές που έγιναν, όπως το λέτε κι εσείς, υπάρχουν μπροστά στην κυβέρνηση, η οποία θα δώσει συνέχεια. Και η Εθνική Συνέλευση ακριβώς αυτό το ρόλο έχει. Θα φροντίσει να υπάρξει συνέχεια στην έκθεση αυτή και να μην υπάρχει πια ετοιμορρησία στη χώρα. Βέβαια, ακόμα και η διεθνής ε, δικαιοσύνη που έχει περισσότερα μέσα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δηλαδή, που έχει πολύ περισσότερα μέσα από την ακτή του, ε, δεν έχει τελειώσει με τον προηγούμενο πρόεδρο της χώρας, ε, το κατηγορητήριο δηλαδή δεν είναι ακόμα πλήρες. Άρα χρειάζεται χρόνος πρώτα να φτιαχτεί η δικαιοσύνη και μετά σιγά σιγά να αρχίσει να λειτουργεί. Χρειάζεται λοιπόν να οικοδομηθούν οι θεσμοί γι' αυτό και δεν είχαμε χρόνο. Τώρα που αρχίζει να λειτουργεί κανονικά πλέον το κράτος, τώρα αρχίζουμε να ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, όπως αυτά που αναφέρει η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστία και όχι μόνο, γιατί εσείς διαβάσατε αυτή την έκθεση, αλλά αν διαβάσετε και την έκθεση της Επιτροπής για την Συμφιλίωση, θα δείτε και εκεί αναφέρονται φοβερά πράγματα, φοβέρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων την εποχή του πολέμου στη χώρα. Αλλά εδώ πρέπει να χαιρετήσουμε την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ακριβώς γιατί εμείς δεν είμαστε όπως η προηγούμενη κυβέρνηση. Να βάλουμε δηλαδή στο σιρτάρι και να την ξεχάσουμε την έκθεση, όχι, τη δημοσίευσαμε στο διαδίκτυο, γιατί θέλουμε οι κάτοικοι τη ακτή ελεφαντοστού να έρθουν αντιμέτωποι με τα εγκλήματα που έγιναν στη χώρα. Εμεί θέλουμε διαφάνεια στη δικαιοσύνη. Θέλουμε δικαιοσύνη να μπορεί να κάνει τη δουλειά τη. Αυτό είναι το τίμημα. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να δώσουμε τη δημοκρατία στη χώρα μα. Και έχουμε αναλάβει αυτό το καθήκον. Τώρα, όλοι όσοι αναφέρονται στην έκθεση αυτή, θα αναλάβουν τι ευθύνε του. Στη δικαιοσύνη. Απέναντι στη δικαιοσύνη. Και για να έρθω σε μια άλλη ερώτηση, εμεί δεν καταλαβαίνουμε πώ είναι δυνατόν ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο επίση θέλει να οικοδομήσει τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου στη χώρα, πώ είναι δυνατόν να βάζει σαν προπόθεση για τη συμμετοχή του στις εκλογέ στη χώρα την ίδια, να βάζει σαν προπόθεση λοιπόν την διακοπή μια δικαστική διαδικασία. Μας λένε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πρέπει να ελευθερώσει τον κύριο Κμπακμπό, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια του. Και μόνο τότε το πολιτικό του κόμμα θα συμμετάσχει στην πολιτική ζωή της χώρας. Μα καταλαβαίνετε που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Η κυβέρνηση λοιπόν της ακτής ελεφαντοστού και το κοινοβούλιο δεν είμαστε σε θέση εμείς να ζητήσουμε από τη διεθνή δικαιοσύνη να ελευθερώσει τον κύριο Γκμπακμπό τη στιγμή που εκείνη είχε αναλάβει ε, την ε, διαδικασία αυτή. Δεν μπορεί εμείς να κάνουμε τέτοια παρεμβολή. Εμείς συμφωνούμε να συνεχιστεί ο διάλογος. Και τον θέλει η κυβέρνηση, τον ζητά. Ήμουν πρωθυπουργό όταν ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μου ζήτησε, προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση τη 1η Ιουνίου του 2011, να μιλήσω με το FPI, με το κύριο δηλαδή κόμμα τη αντιπολίτευση, του οποίου ο πρόεδρο ήταν στη Χάγη και ο οποίο ευθύνεται για ορισμένα εγκλήματα που έγιναν στη χώρα. Παρ' όλα αυτά μου είπαν να συζητήσω μαζί τους για να έρθω στην κυβέρνηση. Αρνήθηκαν όμως. Όσον αφορά τις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές, όταν ο ΙΕ επιβεβαίωσε ότι όλα πήγαν καλά, βάσει κριτηρίων δημοκρατικών διεθνών, τότε μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο οι εκλογές έγιναν με διαφάνεια ή όχι. Οι εκλογές λοιπόν αυτές που οδήγησαν στην Εθνική Συνέλευση πήραν αυτό το κατά κάποιο τρόπο πιστοποιητικό από τον κύριο Μπακιμούν, τον γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί είπανε ότι όντως η διαδικασία έγινε με διαφάνεια, ήταν δημοκρατική, αντιπροσωπευτική για όλον το λαό της χώρας. Συνεπώς, πιστεύω σήμερα ότι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση της ακτής ελεφαντοστού να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να πάει προς την κατεύθυνση του διαλόγου, αλλά και, και πρέπει να πούν ποιος έχει την ευθύνη, που είναι η αντιπολίτευση η οποία δεν συμμετέχει στη δημοκρατική διαδικασία και πρέπει να ζητήσει από την αντιπολίτευση να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία. Είναι σημαντικό. Για την τελευταία ερώτηση. Με ρωτήσατε τι πολιτικές ακολουθούμε για την απάλληψη της ένδυας. Είχαμε 20 χρόνια πόλεμο. Ο μισός πληθυσμός το 2009 ήταν σε ένδυα, 50%. Μετά την κρίση, μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση ανέλαβε μεταρρυθμίσεις. Και αυτό προκειμένου να μπούμε και πάλι στην ανάπτυξη. Για ένα χρόνο είχαμε ανάπτυξη. Νομίζετε ότι φτάνει για να φτάσει ο πλούτος στον κάθε πολίτη. Όχι, η ανάπτυξη αυτή πρέπει να συνεχιστεί πολλά χρόνια για να μπορέσει να έχει και αντίκτυπο και να μειωθεί ο δείκτης ένδυα στη χώρα. Γι' αυτό και λέω και επιμένω και σε εσά αγαπητοί ευρωβουλευτές, η ακτή ελεφαντοστού είναι αλήθεια, βγαίνει από μια κρίση, αλλά συνεχίζει να είναι ευάλωτη. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε τη στήριξή σας, την αλληλεγγύη σας, προκειμένου να παγιωθεί το ποσοστό ανάπτυξης αυτό στην ακτή ελεφαντοστού και έτσι να έχουμε πολλά χρόνια δημιουργίας πλούτου και αυτός πλέον να μπορεί να καταλήξει στον κόσμο και να μειωθεί το ποσοστό ένδυας. Φυσικά, για να απαντήσω στον Ευρωβουλευτή, η Εθνική Συνέλευση έχει ψηφίσει το Εθνικό Τετραετές Σχέδιο Ανάπτυξης που πάει μέχρι το 2016. Προτεραιότητα στο πρόγραμμα αυτό είναι δύο πράγματα. Η εκπαίδευση και η υγεία. Γιατί το γνωρίζουμε ότι για τις υπονάπτυξη χώρες ο πλούτος κατά προτεραιότητα πρέπει να πάει στους πιο ευαίσθητους τομείς. Τα θετικά από την προτεραιότητα αυτή τα επενθύμησε και η Πρόεδρος, ότι δηλαδή στον τομέα της υγείας έχουν γίνει τεράστια βήματα. Δωρεάν περίθαλψη. Πολύ συγκεκριμένα, ας πούμε, είπαμε, οι γυναίκες που περιμένουν παιδί, που είναι σε ενδιαφέρουσα. Αυτές πιο εύκολα μπορούν να έχουν δωρεάν ε, περίθαλψη ή για κάποιες θεραπείες. Είπαμε ότι θα επιτρέψουμε στον πληθυσμό που έχει πληγεί από τον πόλεμο να μπορεί να έχει περίθαλψη δωρεάν. Επίσης, είναι δωρεάν η πρόσβαση στα σχολεία, στο δημοτικό. Το κράτος δηλαδή αγοράζει για τα παιδιά τα βασικά του υλικά και έτσι οι πιο φτωχές οικογένειες που δεν μπορούν να αγοράσουν τα βιβλία, τα τράδια κτλ. Εμείς το κράτος τα αγοράζει και τους τα δίνει δωρεάν. Έτσι το σχολείο γίνεται δωρεάν μέχρι την έκτη δημοτικού. Να λοιπόν κάποια παραδείγματα που έχω να σας δώσω. Κυρία Πρόεδρε, περιμένω το δεύτερο γύρο ερωτήσεων, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. κύριε κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να θέσω μια ερώτηση. Ευχαριστώντας τον Πρόεδρο για τα λόγια του τα τόσο ενδιαφέροντα που μας επιτρέπει να κρίνουμε καλύτερα την κατάσταση που υπηρετεί στην ε, ακτή του ελεφαντοστού σήμερα. Μας ε, επηρεάζουν οι καταστάσεις ε, εκτός Ευρωπαϊκής, της χώρα σας, διότι παλιά το κράτος σας ήταν ναι, το διαμάντι της ε, επιτυχίας. Εμείς ε, είδαμε τον ε, άνοδο αλλά και την πτώση της χώρας αυτής. Μια χώρα λοιπόν που είχε γνωρίσει μια τόσο μεγάλη ανάπτυξη στο παρελθόν, πώς μπορεί μέσα σε τόσο λίγα χρόνια να πέσει τόσο χαμηλά. Ποια είναι λοιπόν η διάρκεια των επιτυχιών ε, και τολμώ να ελπίζω πως ε, ε, η πρόοδος την οποία αναφερθήκατε θα είναι διαρκής, θα είναι βιώσιμη, ίσως να ασφάλω. Σε ό,τι αφορά ανθρώπινα δικαιώματα έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη προχωράει διότι αυτό είναι απαραίτητο, απαραίτητο στοιχείο σε μια ε, δυναμική από την δημοσιογραφική πλευρά χώρα και μπορέσετε να αποκαταστήσετε την ηρεμία και την ειρήνη στην χώρα σας. Βλέποντας τα πράγματα απ' έξω και από αυτούς που κρίνουν την εσωτερική κατάσταση όντας εκτός της χώρας, και αν μπορείτε να με βεβαιώσετε την πληροφορία μας, είναι γεγονό ότι η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης που πριν από την κρίση ε, βρισκόταν στο Αμπιτζάν, ήταν εγκαριστημένη στο Αμπιτζάν, ε, μετάφερε την έδρα της στην Τινησία και είναι έτοιμη να επιστρέψει στο Αμπιτζάν. Εάν αυτό είναι μια πραγματικότητα, τότε αυτό θα έχει μεγάλη σημασία για την χώρα σας ε, Λοιπόν, αυτή η πληροφορία είναι σωστή και πότε πιστεύετε ότι θα μπορείτε να υποδεχτείτε εκ νέου την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης που είναι ε, ένας τουλάχιστον θεσμός που μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανοικοδόμηση της ε, οικονομίας σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόησερ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Σόρο, νομίζω ότι μας περιγράψατε αναλυτικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σας και είπατε ότι η χώρα σας βρίσκεται ε, σε καλό δρόμο, το δείχνει αυτό η επίσκεψή σας εδώ, αλλά και η συνεργασία της χώρας σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσατε για τη διαδικασία συμφιλίωσης. Η ερώτησή μου σε τι βαθμό η διαδικασία συμφιλίωσης υποστηρίζεται από την Αφρική Ένωση καθώς και από την Ένωση χωρών της Δυτικής Αφρικής, διότι φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ να παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά πρώτα καλείται η ε, Αφρικανική Ένωση και οι χώρες της Δυτικής Αφρικής. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προβλέπει να διατεθούν ε, για ε, τη χώρα σας 200 εκατομμύρια ευρώ και με το ενδέκατο πλαίσιο ε, ε, προβλέπεται διπλασιασμός, δηλαδή στα 500 ε, εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την παροχή ενέργειας, θέλετε να ακολουθήσετε νέες οδούς. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πώς προβλέπετε ενίσχυση των μικρών γεωργών και τι ρόλο προβλέπετε για τις γυναίκες ε, στην ε, ανάπτυξη. Και όσον αφορά την ενέργεια και την πρόσβαση στην ενέργεια, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ε, τονίζουμε ότι χωρίς πρόσβαση στην ενέργεια είναι πολύ δύσκολη η ανάπτυξη. Πώς, βλέπ... πώς διαμορφώνεται η δική σας πολιτική ενέργειας. Στα σχέδια σας για την ενέργεια προβλέπετε ε, την περιφερειοποίηση προβλέπετε ε, να υπάρχει γενική πρόσβαση στην ε, ενέργεια. Ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον εαυτό μου. Ε, θυμόμαστε όλοι το δράμα, τη τραγωδία της Μπουκουάλα, το πλοίο που είχε αναβλώσει πήγε στη Φαγέρα με σημαία κάτω χωρών το οποίο μετέφερε παρανόμως ε, τοξικής φύσης ε, εμπορεύματα προς τη χώρα σας. Θυμόμαστε ότι υπήρξαν κάποιοι νεκροί και 20.000 τραυματίες. Επίσης, ε, και η ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω είναι εάν σήμερα τα θύματα αποζημιώθηκαν για τα τραύματά τους που βρίσκεστε σε ό,τι φορά την κάλυψη των ποσών που προέκυψαν μετά αυτό το ατύχημα που ανήρχονται σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Έχετε το λόγο, Πρόεδρε, για να απαντήσετε στο σύνολο των ερωτήσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απαντώντας την πρώτη ερώτηση, εάν η τράπεζα θα επανέλθει στην αρχή του Αλβαριστού, σας διαβεβαιώνω πως η αρχή για την επιστροφή της τράπεζας στην ακτή του είναι κάτι το κεκτημένο. Ε, συζητάμε και ε, συζητάμε και συμφωνούμε τους τρόπους ε, επανεγκατάστασης ε, με τους υπεύθυνους της τραπέζας. Ξεκινήσαμε εναυλώνοντας ένα, μάλλον ένα κτίριο το οποίο θα, στο οποίο θα εγκατασταθεί η τράπεζα. Αυτή είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια επιβεβαίωση των όσων είπα προηγούμενα, να πω δηλαδή ότι το ζήτημα της ασφάλειας στην ακτή του ελευθερωστού σημαντικά έχει βελτιωθεί. Και αυτό δεν είναι μια ανακάλυψη ούτε της κυβερνήσεώς μας, ούτε της ε, ε, Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης. Ας δούμε, πέρασαμε από τον δίκτυ 4 στον δίκτυ 1 κάτι το οποίο δείχνει πως οι διεθνείς οργανώσεις ε, μπορούν να εγκατασταθούν πλέον στις, ε, στην αυτή του όλες οι πρεσβείες ε, επέστρεψαν και όσε δεν το έχουν πράξει έχουν ξεκινήσει την διαδικασία. Πάντως σύντομα θα επανέλθει και η τράπεζα της Αφρικαν... η ανάπτυξη της Αφρικής στο παρελθόν υπήρξαν, ε, υπήρξε συνδυασμό πολλών προβλημάτων που οδήγησε στην κρίση που όλοι γνωρίζουμε. Δεν ε, ήταν ε, κάτι το παράδοξο. Όταν κάποια κρίση πλήττει μια χώρα υπάρχουν κάποια συναισθήματα που αναπτύσσονται ε, θεωρείται ότι έρχονται ξένοι για να πάρουν τις δουλειές των αυτοχθόνων πληθυσμών και ούτω καθεξής και, και όλα αυτά οδηγούν σε μια εχθρότητα, σε ένα μίσος φιλετικό και οι δομές αποδυναμώνονται με τέτοιου είδους κρίσεις και αυτό έζησε και η αρχιευτή του Ελεφαριστού μετά από την μείωση, την πτώση των τιμών πρώτων υλών και αυτό είχε επιπτώσεις ε, επί του συνόλου της επικράτειας. Ε, αρκούσε λοιπόν ε, μια, μια σπίθα για να πάρει φωτιά το όλο οικοδόμημα. Εμεί τώρα οικοδομούμε τον κράτος δικαίου και την δημοκρατία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συναισθήματα που κατέστρεψαν την χώρα μας. Γι' αυτό επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει, να οθήσει την ακτή του εργοδοστού προ την κατεύθυνση του κράτου δικαίου, τη δημοκρατία και του σεβασμού των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Τώρα, για το ζήτημα της διαδικασίας της θα πρέπει να δούμε τη διαδικασία αυτή μια άποψη δυναμική και όχι στατική. Είπα ότι συστήσαμε μια ομάδα ε, εργασίας ε, για την αλήθεια και τη συμφιλίωση. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει πως συμφωνούμε να συγχωρέσουμε, αλλά χρειάζεται η πραγματικότητα επί των ιδεχθών εγκλημάτων που πραγματοποιήθηκαν να γνωστοποιηθεί. Και όσοι πρόκειται να μεταμελήσουν, ας μεταμελήσουν. Και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό συνέβη στην Νότια Αφρική, πιστεύω ότι θα συμβεί και στην ακτή του του. Ήταν ε, σωστό που έγινε στη Ρουάντα όπου υπήρξαν ένα εκατομμύριο θύματα αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και στην ακτή του Λεβαντοστού. Άρα μην νομίζετε ότι αυτό γίνεται με ένα μαγικό ραβδί, από τη μία μέρα στην άλλη όλα σβήνονται, είναι μια πρόκληση. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, θα επιμείνουμε παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν αυτό δεν ε, χάνω την μου, όλοι την εμπιστοσύνη μου. Όλοι λοιπόν ε, πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ε, δουν το συμφέρον του έθνους που δεν ε, εστιάζεται σε έναν ηγέτη αλλά στην ακτή του ελεφαντοστού τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν κρίνω ότι κάθε κόμμα έχει ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβει σε αυτή τη διαδικασία συμφιλίωσης. Και πρόεδρε, εγώ με τα χαράς ε, θα συναντήσω στο Αμπιτζάν ευρωβουλευτές ε, που θα έχουν έρθει στην του Λιπαραστού για να μιλήσουν με την κυβέρνηση διότι έχουν, φέρουν πολλές ευθύνες προκειμένου να προχωρήσουν τα πράγματα, να οθήσουν την διαδικασία της συμφιλίωσης, αλλά και να μιλήσουν και με την αντιπολίτευση και να τους πούν ότι φέρουν ευθύνες και ποιες είναι αυτές. Διότι συχνότατα ε, οι άνθρωποι έχουν το συνέστημα πως όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση όλα είναι σωστά, το είναι απόλυτη αλήθεια κατέχει αντιπολίτευση. Όχι, δεν έχουν έτσι τα πράγματα, μπορεί κανείς να ανοίγει στην αντιπολίτευση και να ασφάλει. Όπως μπορεί να είναι στην εξουσία και να έχει δίκιο. Θεωρώ λοιπόν πως πάνω σε αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας. Τώρα, σε ό,τι τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλήσατε αντίγο παρέθεση και ξέρετε ότι είμαστε μια χώρα ανεξάρτητη από το 1960. Έχουμε σαφή προσανατολισμό. Ξέρετε ότι ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας βάσει την ανάπτυξη της ε, ακτής του και στην ανάπτυξη της ε, Γεωργίας. Αυτή είναι μια απόφαση που λάβαμε τότε, όταν άλλες χώρες επέλεξαν άλλες στρατηγικές ανάπτυξης, τότε ακτή του Ελβανιστού ε, επέλεξε να προωθήσει την ανάπτυξή της μέσω της Γεωργίας. Δουλέψαμε γι' αυτό και επειδή υπήρξα υπουργό άμυνα και πρωθυπουργό απέναντι στο ζήτημα της ανεργίας, όχι μόνο για την χώρα μου, αλλά για όλη την Αφρική. Το πρόβλημα στην Αφρική είναι ένα ζήτημα αφρικανικό. Δηλαδή, έχουμε εκατομμύρια νέους που δεν ε, απασχολούνται, δεν έχουν εργασία, είτε στην Λιβερία, είτε στο Μαλί, είτε στην του Όλοι οι νέοι που πήραν τα όπλα δεν είναι επειδή ότι ένα όπλο είναι ωραίο εμφανισιακά αρέσει στους νέους, αλλά ένα όπλο επιτρέπει σε κάποιους να επιζήσουν, να επιβιώσουν. Γι' αυτό οι νέοι με μεγάλη ευκολία πήραν τα όπλα. Αλλά αυτοί οι νέοι που εξοικειώθηκαν με τον χειρισμό των όπλων θα πρέπει να έχουν μια άλλη συναλλακτική να προτείνουμε κάτι το διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό είναι η εργασία. Σε χώρες λοιπόν όπως η δική μας χώρες υπανάπτυκτες, ποιοι είναι οι κλάδοι που μπορούν να δημιουργήσουν θέσει εργασία για μένα είναι η γεωργία, διότι στη γεωργία δεν έχετε ανάγκη να είστε διπλωματούχος ή να έχετε ένα διδακτορικό για να εργαστείτε. Μπορεί και ένας αναλφάβητο να δουλέψει κάλλιστα στον κλάδο τη γεωργίας. Πιστεύουμε λοιπόν πως για να απορροφηθεί η ανεργία που υπάρχει στη χώρα μας, διότι μιλάμε για 4 εκατομμύρια νέους που κρούν την πόρτα του εργασίας πρέπει να ρίξουμε χρήμα στον τομέα αυτό της, της γεωργίας, διότι το μόνο που θέλουν αυτοί οι νέοι είναι να τραφούν, να τρέψουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τώρα πέρα των ε, καλλιεργιών που είχαμε μέχρι τώρα να αλλάξουμε τις καλλιεργίες μας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και άλλες μορφές γεωργίας. σε ό,τι φορά το θέμα της ενέργειας, αυτό είναι σφαιρικό πρόβλημα. Ναι, οι χώρες μας δεν θα είναι ανταγωνιστικές εάν δεν έχουμε μια πραγματική ικανότητα παραγωγής ενεργειακής, ενεργειακής Ξέρετε ότι η ακτή του δίνει ε, ε, ηλεκτρισμό στην ε, ενέργεια μάλλον στην, ε, στο Μαλί και σε άλλες χώρες. Αν είχαμε όμως δυνατότητα θα δίναμε και στη Λιβερία και στη Σιέρα Λεόνα και σε άλλες. Πρόκειται για ένα ζήτημα λοιπόν πολύ σημαντικό, ζωτική σημασία. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να επιληθεί σε επίπεδο μικρών κρατών. Θα πρέπει να επιληθεί σε περιφερειακό. Υπάρχει η Νιγερία που ε, παράγει ουράνιο και κυρία Πρόεδρε για να μην ξεπεράσω και τον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, ξέρω ότι είναι ιερή η ώρα για εσάς, ενώ στην Αφρική μπορούμε να επιμηκύνουμε τις παρεμβάσεις μας. Ε, θα έλεγα λοιπόν το ζήτημα της ενέργειας είναι ζωντική σημασίας για να καθιστούσουμε τις χώρες της Αφρικής ικανές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της χιλιετίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε της Εθνικής Συνέλευσης της Εκτής Ελεφαντοστού για την επίσκεψή σας και για το ότι μοιραστήκατε μαζί μας την ανάλυση σας για την κατάσταση σήμερα στην χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Oui, c'est ça. Je vais continuer maintenant avec d'autres questions. J'attends une minute parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans la salle.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 Nous allons continuer. Euh. Συνεχίζουμε. Είμαστε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων για την Ελληνική Συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κυριμπάτι. Ο κύριος Νόισερ είναι ο εισηγητής μας. Ξέρουμε ότι η αρμόδια επί της ουσίας Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι η Επιτροπή Αλίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλώς θα συμφωνήσει ή θα διαφωνήσει με το πρωτόκολλο. Συνεπώς, δίνω το λόγο στον κύριο Νόισερ ευθύς αμέσως για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε, αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Αλίας. Εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης γνωμοδοτούμε μετά από πολλές ε, συνομιλίες. Στη γνωμοδότησή μου συστήνω η συμφωνία αλίας με το ε, να μην συμφωνήσουμε με τη συμφωνία αυτή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ε, διαπραγματεύσεις της ε, για τη Συμφωνία Αλίας Ε, δεν έχει λάβει υπόψη την ε, συμφωνία Ναουρού. Ε, διότι προβλέπεται εδώ έλεγχος της αλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συμφωνία με το Κυριμπάτη δεν παίρνει ως βάση τη συμφωνία Ναουρού και δεν προβλέπει το σύστημα ελέγχου για τα σκάφη, το VDS. Ε, έτσι υπονομεύουμε την Περιφερειακή Συμφωνία Αλίας ε, στον Ειρηνικό. Και αυτό βρίσκω ότι είναι λάθος. Εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, στην συνέλευση ΑΚΕ, πάντα κηρύττουμε η περιφερειακή συνεργασία να προωθείται στα, στις χώρες ανάπτυξης, ε, ε, στη, στον ειρηνικό, στον τομέα της Αλίας υπάρχει τέτοια περιφερειακή συμφωνία. Εάν όμως εμείς ε, συνάψουμε συμφωνία με το Κυριμπάτι, υπονομεύουμε αυτήν την ήδη υπάρχουσα περιφερειακή συνεργασία. Γι' αυτό η πρότασή μου προς την Επιτροπή είναι να απορρίψουμε τη συμφωνία υπό τη μορφή που έχει και σύντομα να υποβάλουμε νέα συμφωνία, νέα πρόταση συμφωνίας που να σέβεται την ε, συμφωνία του Ναουρού και να την βελτιώνει. Εάν συμφωνήσουμε με τη Συμφωνία Λία με το Κυριμπάτι υπό τη μορφή που έχει, θα δημιουργήσουμε αρνητικό προηγούμενο, διότι έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ε, υπονομεύσει, ε, θα έχει αγνοήσει μια περιφερειακή συμφωνία. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν απορρίψει την πρόταση αυτή, αυτό οικονομικά δεν θα είναι το τέλος του κόσμου για το Κυριμπάτη. Το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού θα χάσει το Κυριμπάτη. Ε, τέτοιο μερίδιο αντιπροσωπεύει η συμφωνία με το Κυριμπάτη. Αυτή η απώλεια του 1% του προϋπολογισμού θα είναι κάτι το οποίο θα ισχύει μόνο στο διάστημα που θα χρειαστεί το Κυριμπάτι και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψουν νέα συμφωνία με βάση τη Συμφωνία Ναουρού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Μπορώ μόνο να τονίσω τα όσα είπε στα έγγραφα της σημερινής συνεδρίασης. Ε, πέρα από την γνωμοδότηση ε, του κυρίου ε, Νάουζερ, έχουμε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμού που συμφωνεί με τη συμφωνία, αλλά η Επιτροπή αυτή μάλλον έχει λάβει υπόψη μόνο ε, την οικονομική πτυχή. Σημαντική διαφορά δεν υπάρχει με την προηγούμενη συμφωνία, άρα μπορεί η Επιτροπή Προπολογισμού να πει ότι εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εγώ συμφωνώ με τον κύριο Νάουζερ, πρέπει να ακολουθήσουμε τη δική μα πολιτική κατεύθυνση. Όταν ε, λέμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε την ε, συνεργασία ανάμεσα στι αναπτυσσόμενε χώρε, ειλικρινά εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε πώ μπορεί το κυριπάτι να συμφωνήσει με μια τέτοια συμφωνία, διότι έτσι θα αντιμετωπίσει σημαντικέ ε, ε, ε, συγκρούσεις. Πρόκειται λοιπόν για μια μικρή χώρα ε, ΑΚΕ η οποία συνέχεια ε, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ε, αύξησης της στάθμης ε, των ωκεανών. Αλλά εν πάση αυτό δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την ε, γραμμή που πρεσβεύουμε και νομίζω ότι μπορούμε να ξαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία. Η αλία είναι πολύ σημαντική για το Κυριμπάτι, αλλά η συμφωνία αυτή αντιπροσωπεύει μόνο το 1% του υπεροπολογισμού της χώρας. Γι' αυτό συμφωνώ με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Πόγκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Νόιζερ για το έργο του. Όπως γνωρίζετε, ο Ερηνικός είναι μια περιοχή, εντάξει δεν λέω ότι εγώ τη γνωρίζω καλά, αλλά έρχομαι από εκεί. Οπότε κάτι γνωρίζω. Είναι δικιά μου περιοχή. Το Κυριμπάτι είναι πολύ κοντά στην Νέα Χαλιδονία. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τις ανησυχίες του κύριου Νόιζερ για την τήρηση των ε, συμφωνιών που συνάπτει η χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του Κυριμπάμπη στα πλαίσια της Συμφωνίας Ναουρού. Εγώ συμφωνώ με την αρχή αυτή. Όμως από το πρωτόκολλο και από τις ανταλλαγές που είχαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εδώ λυπάμαι βέβαια που δεν είναι παρούσα εδώ σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πάντως θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εμποδίζει το κυριμπάτι να τηρήσει τις διεθνείς του δεσμεύσεις. Εφόσον το επιθυμεί το κυριμπάτι, εφόσον εφαρμοστεί το πρωτόκολλο, θα μπορεί να μεταγράψει το σύστημα του σε VDS, έτσι όπως αναφέρεται στην ίδια τη συμφωνία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ούτε και αυτές στηρούν τον ΠΕΤΕΣ με τις χώρες του ειρηνικού. Αλλά όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στα πλαίσια της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλίας του Ειρηνικού. Με το πρωτόκολλο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει την βιώσιμη αλία, με διαφάνεια. Αυτό απαιτούμε και την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, έχουν γίνει κάποιες εκτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φαίνεται ότι το πρωτόκολλο τηρεί πλήρως τα όσα αναφέρουν οι συμφωνίες του Ναουρού και του Παουρού. Μία ρήτρα αναθεώρησης στο πρωτόκολλο μπορεί να προβλέψει για τις οικονομικές προσαρμογές από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ανάλυση ex post θα έχει σαν αποτέλεσμα το πρωτόκολλο να ωφελήσει και τις δύο πλευρές και να ενισχύσει την ανάπτυξη του Κυριμπάτη. Επ' αυτού λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Κυριμπάτη έχει χαμηλούς πόρους και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του νέου αυτού πρωτοκόλλου δίνει 1.325.000 ευρώ ετησίως, τόσο για την πρόσβαση στους ελευτικούς πόρους, όσο και για να στηρίξει την ελευτική πολιτική του Κυριμπάτη. Για τρία χρόνια δηλαδή 4.428.000 ευρώ. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε βέβαια και τα χρήματα που δίνουν οι πλειοκτήτες. Για μια χώρα λοιπόν η οποία εξαρτάται τόσο πολύ από ελευτικούς πόρους, μιλάμε για 23 με 33% έσοδα για τη χώρα. Πολύ σημαντικό. Επίσης, με το πρωτόκολλο αυτό ενισχύεται η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες του Ειρηνικού. Σε περίπτωση που απορριφθεί το πρωτόκολλο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδυναμώνεται στα πλαίσια του Περιφερειακού Οργανισμού Αλίας του Ειρηνικού προκειμένου να προωθήσουμε δηλαδή τη βιώσιμη αλία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και η Αυστραλία ή ακόμα και η Νέα Ζηλανδία είναι πολύ παρούσες και είναι ικανοποιημένε. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσυρθεί από την περιοχή θα αντικατασταθεί και οι ευρωπαϊκές μας αξίες θα γνωριθούν Πλήρω εξαιτία άλλων οικονομικών συμφερόντων. Υπενθυμίζω επίσης ότι η Επιτροπή μας είχε εγκρίνει το πρωτόκολλο για τη Μικρονησία και τις νήσους του Σολομώντα, ενώ το πρωτόκολλο δεν αναφερόταν στο VDS. Δεν μπορεί να έχουμε δύο διαφορετικές πολιτικές, ανάλογα με το για ποια χώρα πρόκειται, πρέπει να είμαστε συνεπείς. Γι' αυτό και θα υποβάλω τροπολογία ζητώντας την στήριξη του πρωτοκόλου, διότι πιστεύω ότι το διεθνές δίκαιο υπερέχει των άλλων. Ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Ιζαμπέλ Λεβίνη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που άργησα. Δεν άκουσα λοιπόν την παρουσίαση του εισηγητή, δυστυχής, ε, δυστυχώς ε, ούτε άκουσα τις δηλώσεις της Κομισιόν. Αλλά θα ήθελα να πω όμως ε, ότι ως ε, εισηγητής για την ε, συμφωνία ε, με το Κυριμπάτη στην Επιτροπή Αλίας, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Νόιζερ. Από πλευράς ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντικό να θίξουμε τα θέματα που θίγει ο κύριος Νόιζερ στην γνωμοδότησή του για τη Συμφωνία Αλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, Ε, έχει πολύ κακό όνομα στην περιοχή λόγω του τρόπου που διαπραγματεύεται αυτές τις ε, συμφωνίες αλίες. Ε, και κύριε Πόγκα, αυτό αφορά και τις συμφωνίες με τη Μικρονησία και τις νήσου Σολομώντα. Δυστυχώς, όταν διαπραγματευόμασταν την συμφωνία αλίας με τη Μικρονησία στην Επιτροπή Αλίας, αυτό διάφυγε της προσοχής μου. Ε, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται στην άλλη πλευρά του πλανήτη και δεν είναι πάντα εύκολο να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει. Ξέρουμε όμως ότι ε, το Κοινοβούλιο της Μικρονησίας απέρριψε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να αναγνωρίσει ε, το πρόγραμμα VDS καθώς και τη συμφωνία Ναουρού. Ε, και διαπραγματευόταν μόνο οι μέρε ε, σκαφών στη θάλασσα. Το ίδιο, ε, το ίδιο ισχύει για την συμφωνία με τις νήσους Σολομώντα. Και αυτό το έχουμε συζητήσει εκτενώς στην Επιτροπή Αλίας. Η κατάσταση έχει ως εξής. Έχουμε μια σειρά μικρών νήσων κρατών που επιτέλους κάτι όχι πολύ συνηθισμένο, έχουν προχωρήσει πολύ στη συνεργασία μεταξύ τους ε, για τη διαχείριση του βασικού φυσικού πόρου τους. Ε, είναι ο μόνος φυσικός πόρος που μπορούν να έχουν στην περιοχή αυτή, η αλία δηλαδή, και ε, ο πόρος αυτός είναι ιδιαίτερα πολύτιμος εδώ και πολύ καιρό. Ε, τα ε, νησιά αυτά αγωνίζονται να μεγιστοποιήσουν ε, το, το κέρδος τους από την αλληλεία. Και πρόκειται για μοιρασμένα αποθέματα και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούν για τη διαχείριση των αλλιευμάτων αυτών. Και η Συμφωνία Ναορού επιδιώκει Εάν ένα ε, απόθεμα ε, ε, περνάει τον ένα χρόνο πάρα πολύ καιρό σε μία περιοχή, ενώ τον επόμενο χρόνο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη άλλου νησιού, να μπορούν να ανταλλάσσουν οι μέρες αλίας και πρόκειται για σημαντική πρόοδο στο μέρος αυτού του κόσμου και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κανένα, κανένας από τους συμβαλόμενους της Συμφωνίας του Ναουρού να μην συμφωνήσει να πουλήσει πιο φτηνά ε, τα αποθέματα από τα άλλα μέλη της Συμφωνίας. και αυτό συνέβη με, την, με τις νήσους Σολομώντα. Ε, πολλούσαν ανατόνο ε, τα αλλιεύματα αυτά με τρόπο που δεν μπορούσαν να δεχτούν τα άλλα ε, συμβαλόμενα μέρη της Συμφωνίας Ναουρού. Και ε, δύο φορές παρευρέθηκα σε ε, περιφερειακές ε, συνεδριάσεις αλίας στην περιοχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά θεωρείται πολύ καλός παράγοντας, διότι ουσιαστικά είμαστε ο βασικός πάροχος αναπτυξιακής βοήθειας και μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής βοήθειας αφορά την αλλήλεια. Όσον αφορά όμως την αλλήλεια δυστυχώς, και ε, σας το εγγυώμαι αυτό, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαφωνήσει. Ε, όσον αφορά την αλληλεία όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ κακή εικόνα στην περιοχή, επειδή οι χώρες διαπιστώνουν ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ε, να παρέμβει και να διαιρέσει τις χώρες ε, διαπραγματευόμενοι με τις χώρες μία-μία και λέγοντας ότι εμείς δεν δεχόμαστε τους όρους της Συμφωνίας Εναουρού, εμείς θέλουμε να αγοράσουμε ε, τα, τα αποθέματα αυτά ε, ε, με τους όρους που θέλουμε εμείς. Κάτι που δημιουργεί τεράστιες συγκρούσεις και ένταση ανάμεσα στα νησιά κράτη του Ειρηνικού. Και αυτό είναι το κλειδί, αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα να, καθοριστεί, ε, να καθοριστούν τα σημεία αναφοράς για το VDS, πόσα ε, ψάρια αλλιεύονται κάθε μέρα. Ξέρω όμως ότι επίσης στην περίπτωση του Κυριμπάτη ε, έγινε μια τεχνική συνάντηση, μια συνάντηση τεχνικής ομάδας των συμβαλωμένων της Συμφωνίας του Ναουρού, όπου διαπιστώθηκε ότι το Κυριμπάτι ξεπερνάει τις μέρες αλληλείας του που δικαιούται. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά ήταν σημαντική υπέρβαση, νομίζω κατά 30 ή 40% παραπάνω από ε, τις ε, ημέρες ε, που ε, είχαν δοθεί στο Κυριμπάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης αλλιεύει στην περιοχή αυτή και φαίνεται ότι η αλλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μετατρέπεται σε μέρες αλληλείας προστίθεται δηλαδή σε αυτές τις μέρες ε, οι μέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα και αν ε, συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία με το Κυριμπάτι, το Κυριμπάτι υπερβαίνει το, τις μέρες που δικαιούται. Πάρα πολύ σημαντικό είναι λοιπόν η Επιτροπή Ανάπτυξης να συνεχίσει να τονίζει και να επικρίνει και να τονίζει ότι εμεί θέλουμε να προωθήσουμε την ε, περιφερειακή συνεργασία ε, ανάμεσα στι αναπτυσσόμενες χώρε. Και ε, αντί να πούμε ότι, α, κοιτάξτε, εμεί δεν τεχόμαστε τις μεταξύ σα συμφωνίε, εμεί θέλουμε να διαπραγματευτούμε μαζί σας με τον καθένα από εσά ξεχωριστά, αυτό είναι το πρόβλημα. Και ξέρω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πιστεύει και συμφωνώ. Θα ήταν ατυχές η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει θέση στην ε, περιφερειακή οργάνωση αλληλείας, αλλά δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική αγορά για τον τόνο της, του ειρηνικού. Ε, ο ειρηνικός ε, παράγει το 40% της, παραγωγής, της παγκόσμιας παραγωγής τόνου και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός αγοραστής. πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό που λέμε εμείς θα βελτιώσει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. αντί, το, αντί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιπροσωπεύει τέσσερα σκάφη, διότι μιλάμε για πολύ λίγα σκάφη που αλλιεύουν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας του Κυριμπάτη. Δεν έχω καμία αντίρρηση να βρίσκονται εκεί τα σκάφη μας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε την συμφωνία ώστε να βρίσκεται στα πλαίσια της βιώσιμης αλληλείας, να μην ε, ε, βρίσκεται έξω, να, να, μην ε, εξαιρείται από τις μέρες που, ε, ε, αποδίδονται στο κυριπάτι και δεν θέλουμε ε, να πληρώνουμε ε, άλλη τιμή από αυτήν των μικρών κρατών νήσων και τα μικρά νησιά αυτά θέλουν να αυξήσουν το σημείο αναφοράς και το Κυριμπάτι ήταν ε, το μόνο κράτος που δεν ήθελε να αυξήσει την παρούσα τιμή που είναι 400-500 δολάρια την ημέρα. 4.000-5.000 ε, ε, δολάρια την ημέρα, συγγνώμη. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά πληρώνει λιγότερα πόσα όσα θα έπρεπε με τη συμφωνία αυτή. Άκουσα να λέγεται κάτι για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, ξέρω ότι η Ιαπωνία Μάλλον δεν είμαι βέβαιη για το, όσον αφορά τη Ιαπωνία, αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε διαπραγματεύονται νέα περιφερειακή συμφωνία υπό τους όρους του VDS. Δεν επιμένει λοιπόν πάνω σε κάτι διαφορετικά. Α, να τα νούμερα. Λοιπόν, το Κυριμπάτι εξεπέρασε σχεδόν κατά 100% ε, τις ε, ημέρες ε, που το αποδόθηκαν. Το ποσοστό λοιπόν είναι πολύ υψηλότερο από το 30% όπω σας είπα εγώ. Και κατά βάση, εάν κατακαιρματίσουμε αυτή τη συνεργασία, αυτό θα σημάνει σημαντική οικονομική απώλεια για όλες τις χώρες αυτές, διότι εάν δεν συνεργάζονται μεταξύ τους, τότε δεν θα ελέγχουν τους φυσικούς τους πόρους κάτι καταστροφικό για όλη την περιφέρεια και κάτι που δεν συνάδει με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κορέα και η Ιαπωνία επίσης εφαρμόζουν το σύστημα VDS. στις ε, συμφωνίες ε, στην περιοχή, όπως και η Κίνα και η Νέα Ζηλανδία. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη μεγάλη δύναμη που δεν δέχεται τους όρους αυτούς. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διορθωθεί. Συμφωνώ με την ε, Κομισιόν ότι χρειαζόμαστε ε, διαφάνεια, αλλά τα αποθέματα αυτά φαίνονται να βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση και θα πρέπει να επιτρέψουμε στην περιφέρεια αυτή να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ όλους και όλες σας. Δεν εκπροσωπείται η Κομισιόν για τα θέματα της Αλίας να προσθέσω και εγώ στη, την άποψή μου στα όσα είπατε είμαι κατά <clears throat> αυτής της συμφωνίας αυτής και προτείνω να την καταψηφίσουμε η ψηφοφορία θα διεξαρθεί στην συγγνώμη στον κύριο Νόουσερ να δώσω το λόγο καταρχήν για να ολοκληρώσω και μετά Κύρια Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι η κυρία Λεβέν ε, ανέφερε αναλυτικά το πρόβλημα, περιγράψε αναλυτικά το, πρόβλημα από πλευράς της Επιτροπής Αλίας. Ε, δεν θα αναφερθώ σε αυτήν την πτυχή, αλλά να τονίσω τις, τις αναπτυξιακές πτυχές. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε εταίρος που να ε, οδηγήσει σε κατακαιρματισμό στην περιοχή ε, και καταστροφή της περιφερικής συνεργασίας. Δεν είναι αυτή η θέση της Επιτροπής μας. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε να μην έχουμε ε, απομονωμένες συμφωνίες με την κάθε χώρα, αλλά να πληρούμε τους όρους της Συμφωνίας Ναουρού. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή ε, τροπολογιών είναι η 3η Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι και ψηφίζουμε στις 24. Περνάμε τώρα στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης που είναι ο συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014 με 2020. Ο συνδυασμό αυτός, αλλιώς blending, είναι ένα επίκαιρο θέμα για την καινοτομία όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μια σημαντική αύξηση των ποσών που πηγαίνουν ε, για το λόγο αυτό στα διάφορα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης. Από την άλλη, η πλατφόρμα εμπειρογνωμένων που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2012 για να μάθει περισσότερα πράγματα όσον αφορά τον συνδυασμό αυτό και, οι βελτιώσεις που, και για τις βελτιώσεις που έχουν γίνει ολοκληρώνει τις εργασίες της. Οπότε τώρα θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα και θα τα συζητήσουμε στην Επιτροπή μας. Εξαιτία τη μείωση τώρα της, ε, του προπολογισμού για την αυτοξιακή βοήθεια και για να στηρίξουμε τις πολιτικές προτεραιότητες, οι δανειστέ ε, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και τη γνώση του ιδιωτικού τομέα στο θέμα της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη. Ο συνδυασμό έχει να κάνει κυρίως με έναν μηχανισμό που φτιάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνδυάσει την δημόσια βοήθεια με ε, δάνεια από ε, πιστώσει από δάνεια από τον ιδιωτικό τομέα ή από εμπορικές επενδύσεις ακόμα. Θα ακούσουμε πρώτα τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εκπώνησαν την μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή μας για τις δυνατότητες που προσφέρει ο συνδυασμός αυτός, αλλά και για τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό το μέσον. Ο κύριος Μπαρτ Στάς, που είναι εισηγητής μας επιμονή μου βάσεως για τον συνδυασμό αυτών, αλλά και παρατηρητής από πλευρά της Επιτροπής μας στα πλαίσια της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον συνδυασμό των ε, δανείων και της χρηματοδότησης, θα μας παρουσιάσει την άποψή του και τους προσανατολισμούς που φαίνεται να καταλήγει η προβληματική αυτή. Θα δώσω όμως το λόγο πρώτα στον κύριο Πέντρο Μωραθάν, που είναι και ο συντάκτης της μελέτης. Έχει το λόγο για 15 λεπτά το πολύ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συνδυασμένη χρηματοδότηση στην πράξη έχει δείξει αυτό που λέμε και εμείς στην μελέτη μας, ότι δηλαδή έχει θετικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, συνδυάζεται η δημόσια χρηματοδότηση με εκείνη από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, επιτρέπεται η χρηματοδότηση μακροχρόνιων προγραμμάτων που αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν να χρηματοδοτηθούν αν δεν γινόταν αυτός ο συνδυασμός. Τρίτον, καταδεικνύει η μελέτη μας επίσης ότι μπορούν να προσθεθούν και άλλες συνεισφορές από τα κράτη-μέλη και επίσης ενισχύεται και η ορατότητα η προβολή δηλαδή των δράσεων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ανάπτυξης. Με τη δημιουργία της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μέρη χρηματοδότηση στον τομέα της εξωτερικής συνεργασίας του Δεκεμβρίου του 2012, δώσαμε ένα βήμα σημαντικό προς τα μπρος για την παγίωση των μηχανισμών που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Κατά τη γνώμη μας, η δημιουργία της πλατφόρμας αυτής ανοίγει νέες δυνατότητες για να καθοριστούν προϋποθέσεις και προδιαγραφές όπως επίσης και στρατηγικές που επιτρέπουν να βελτιώσουμε όχι μόνο την ποσότητα της χρηματοδότησης, αλλά και πάνω απ' όλα την ποιότητα. Με την προοπτική αυτή λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να δούμε την δομή της προτινόμενης διακυβέρνησης μέσα στην πλατφόρμα αυτή, που συνδυάζει μία ε, πολιτική ομάδα η οποία θα ασχολείται πιο πολύ με την πολιτική κατεύθυνση δηλαδή, αλλά ε, συγχρόνως συνδυάζεται αυτό και μία τεχνική ομάδα που θα ασχοληθεί πιο πολύ με την εφαρμογή. Πρόκειται δηλαδή, η πλατφόρμα αυτή είναι ένα φόρουμ που έχει ως αποστολή να συνδέει όλα τα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον πολιτικό τομέα και στον τεχνικό υπέρ της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της, του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας. Τώρα, προκειμένου να βελτιωθεί η δομή της διακυβέρνησης των διάφορων περιφερειακών μηχανισμών που έχουμε από το 2007 και μετά, εδώ θέλουμε να πετύχουμε καλύτερη συνοχή ανάμεσα στους διάφορους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στους περιφερειακούς μηχανισμούς και ε, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα των κρατών μελών. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία βάση των εργασιών των δύο ομάδων. Και εδώ θέλω να τονίσω τις εξής πτυχές που αναφέρονται και στην μελέτη μας. Πρώτον, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη δομή διακυβέρνηση των διάφορων περιφερειακών μηχανισμών, ιδιαίτερα όσον αφορά την συμμετοχή των δικαιούχων. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλους τους μηχανισμούς κάνει ένα καλό σχεδιασμό και επιτρέπει να εντοπιστεί κάποιος υπεύθυνο πολιτικά που θα εφαρμόζει την στρατηγική που έχει να κάνει με την απάλληψη της έδνοιας. Έτσι όπως ορίζονται οι στόχοι αυτοί στη Λισαβόνα. Έπειτα πρέπει να διευκρινίσουμε διάφορα στοιχεία που έχουν να κάνουν με σύγκρουση συμφερόντων. Κυρίως υπάρχει ο μηχανισμός του ETF στην Αφρική. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αντίληψη στον κόσμο, στην κοινωνία των πολιτών, ότι η Προεδρία της Τεχνικής Ομάδας μπορεί να επηρέασει πάρα πολύ το γενικό προσανατολισμό των προγραμμάτων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί παρετέρω. Στη μελέτη μας συστήνουμε εμείς να υπάρξουν σαφείς και κανόνες με διαφάνεια που να επιτρέπουν και εξάντε και εξπόστε την εκτίμηση του κατά πόσο οι μηχανισμοί που χρηματοδοτούνται από την επίσημη συνεργασία του ΜΠΟΤΑ ανταποκρίνονται στην πολιτική την αναπτυξιακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα η ανάλυση που γίνεται των δομών διακυβέρνησης πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και την προοπτική ακριβώ αυτή της καταπολέμησης της ένδυας. Άρα πρέπει να αναλύεται σε τι βαθμό οι μηχανισμοί, που λαμβάνουν, οι μηχανισμοί υπόψη τα συμφέροντα και τις ανησυχίες των ομάδων στόχος. Οι περιφερειακοί μηχανισμοί προς το παρόν δεν έχουν ανοίξει πλήρως την πόρτα στην συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και δεν έχουν πετύχει να διευκρινίσουν, να καθισκάσουν μάλλον πλήρως τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό φαίνεται από την κυβερνητική δομή των ε, μηχανισμών που είναι από πάνω προς τα κάτω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εκπροσωπείται ιδιαίτερα στη συντονιστική επιτροπή της πλατφόρμας, έτσι ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης ώστε να αλλάξει η αντίληψη αυτή που υπάρχει μέχρι τώρα στον κόσμο. Όσον αφορά τώρα τον ε, προσανατολισμό για την απάλληψη της ένδυας. Εδώ πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχουν οι υπάρχοντες περιφερειακοί μηχανισμοί. Έτσι θα εξαφανιζόντουσαν πολλές αμφιβολίες. Άρα να δούμε πώς συνεισφέρουν οι μηχανισμοί συνδυασμένων χρηματοδοτήσεων, blending, σε σχέση με τους στόχους της χιλιετίας. Επιπλέον πρέπει να γίνει και μια ανάλυση για το τι συμφέρει την ε, χώρα εταίρο. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη βέβαια τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο CSP, δηλαδή στα έγγραφα για τη στρατηγική της κάθε χώρας. Έπειτα η ανάλυση να γίνεται και για την ποσότητα αλλά και για την ποιότητα της βοήθειας και να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνία των πολιτών. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να εξισορροπηθεί έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα των επιπτώσεων των μηχανισμών αλλά συγχρόνως να βλέπουμε και πώς οι δικαιούχοι αντιλαμβάνονται την βοήθεια αυτή. Η ανάλυση των επιπτώσεων δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο φαινόμενο της μόχλευσης, δηλαδή στο πόσο μεγαλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Πρέπει να αξιολογείται πάντα η ποιότητα και κυρίως πόσο βιώσιμη είναι πόσο βιώσιμες είναι οι αλλαγές που γίνονται. Και βάσει μιας τέτοιας ανάλυσης πρέπει να χρησιμοποιούμε και έναν πολυδιάστατο ορισμό για την ένδια, όπως έχουμε κοινών από το ΕΣΕΒΕ. Πρέπει να γίνεται και ανάλυση κινδύνων. Όσον αφορά τώρα το ρόλο των διαφόρων φορέων, εμείς πιστεύουμε ότι εδώ υπάρχει μια ευκαιρία να βελτιωθεί η συνεργασία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δουλέψουμε βάσει των μηχανισμών συντονισμού, έτσι όπως καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως βάσει του κώδικα διοντολογίας. Άρα, όπως ακριβώς το λέει και η πλατφόρμα, ο ρόλος ε, συντονιστικός δεν μπορεί να ανατίθεται σε ένα μόνο όργανο, στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για παράδειγμα. Επίσης, αν ο στόχος είναι να κινητοποιήσουμε επιπλέον πόρους από τις χώρες μέλη, τότε η πλατφόρμες και οι μηχανισμοί πρέπει να διέπονται από ευελιξία. Όσον αφορά τώρα το facing out, την διαφοροποίηση, η λειτουργία δηλαδή των μηχανισμών αυτών όταν πρόκειται για χώρες μεσαίων εισοδημάτων ή χαμηλών εισοδημάτων, όταν πρόκειται για μεσαία εισοδήματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι της χρηματοδότησης, γιατί όπως λέμε και στην μελέτη μας, Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι υπερχρέωσης που πρέπει να διαχειριστούμε ε, βάσει των κανόνων διαχείρισης ε, χρέους. Όπως επίσης και το θέμα της μόχλευσης που λέγαμε πριν και αυτό πρέπει να λυθεί υπόψη και πώς θα προχωρήσει ο πληθωρισμός μετά από μια τέτοια βοήθεια. Οι χώρες λοιπόν μεσαίων εισοδημάτων και χαμηλών ε, εισοδημάτων δεν πρέπει να εξεταστούν μόνο βάσει των κατακεφαλήν εσόδων. Αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη διεθνή συνεργασία. Το ίδιο ισχύει και για τη συνδεδεμένη στήριξη. Πάντως η ίδια η λογική των μηχανισμών έχει σαν αποτέλεσμα να ελοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι στην αξιολόγηση του peer review του S&D. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται, αλλά δεν πρέπει να γίνεται με οποιοδήποτε τίμημα. Κάποιες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έθεσαν και κάποιες ερωτήσεις και ανησυχίες προς προβληματισμό και μελέτη που πρέπει να ληφθούν υπόψη αξιολόγησης. Εμείς στη μελέτη μας λέμε ότι ένας τρόπος για να φροντίσουμε για την απάλληψη της ένδυας είναι να γίνεται ανάλυση επιπτώσεων εξάντε όπως έχει αναπτύξει και ο ΣΑ. Πολλές φορές πρόκειται για επενδύσεις σε υποδομές που γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ο προσανατολισμός τους δεν είναι πάντα υπέρ των πιο φτωχών ή δεν τηρούν πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και πρέπει να ελέγχουμε όλες τις διόδους για να αποφασίσουμε ποια είναι τα προγράμματα εκείνα τα οποία θα καταλήξουν καλύτερα σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη στις ομάδες, στόχο δηλαδή. Τα μέσα συνδυασμένης χρηματοδότησης βασίζονται, όπως γνωρίζουμε, στην ε, πρόθεση τελικά του δημοσίου χρέους. Και αυτό συμβαίνει κυρίως στις χώρες μεσαίων εισοδημάτων. Σε περίπτωση αστάθειας των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών, τότε το θέμα του χρέους μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση κινδύνου των μηχανισμών που γίνεται. Είναι σημαντικό επίσης οι μηχανισμοί του συνδυασμένου, της συνδυασμένης χρηματοδότησης να είναι διάφανοι και να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι δείκτες για τη βιωσιμότητα του χρέους και να δούμε τι σχέση έχουν αυτοί οι δείκτες με τα όρια και με τους δείκτες που χρησιμοποιεί το Διεθνές Μεσονατικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζη στην διαδικασία βιωσιμότητας του χρέους. Δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών που έχουν οι χώρες δωρητές και που αναφέρθηκε εδώ, υπάρχει ο κίνδυνος οι μηχανισμοί συνδυασμένης χρηματοδότηση να να περάσουν τις αρμοδιότητες σε άλλους τομείς. Δηλαδή, να υπάρξει τελικά επιπλέον κόστος μπορεί να υπάρξει μια χρηματοδότηση συνδυασμένων χρηματοδοτήσεων με παραπάνω όμως κόστος γιατί επειδή θα υπάρξει μεγαλύτερη απόδοση για τους δωρητές. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται εφόσον θέλουμε να παλύψουμε την ένδια από διάφορες χώρες. Εμείς πιστεύουμε ότι για να αποφευθούν οι κίνδυνοι αυτοί θα έπρεπε να καθοριστούν κώδικες που να καθορίσουν τον προσανατολισμό των προγραμμάτων. Κάτι που κάνουν ορισμένες χώρες μέλη. Αυτό θα ήταν μια διόρθωση που θα γίνεται στα πλαίσια της πλατφόρμας με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει ενός τέτοιου κώδικα θα μπορούσαμε να καθορίσουμε αν ένα πρόγραμμα καταπολεμάει απευθεία την ένδια άμεσα ή το κάνει έμεσα ή σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή αν υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων ή υπάρχει κάποια κοινωνική αδικία ή αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα και τους περιφερειακούς μηχανισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στάση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, είναι καλό που ακούμε ποια είναι η αρχή των συνδυασμένων αυτών χρηματοδοτήσεων. Έχουμε διαβάσει κείμενα, τα οποία εξηγούν πώς λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός και τι αλλαγές γίνονται και πώς ο συνδυασμός αυτός διευκολύνει και το χρέος των χρόνων. Υπάρχει και ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης για την ανάπτυξη. Υπάρχει και συμφωνία συνεργασίας με τους δικαιούχους Υπάρχουν ένα σωρό κείμενα δηλαδή τα οποία εξηγούν το μηχανισμό αυτόν. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο που μας πέρασε, στη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου, ε, υπερψηφίσαμε ένα ψήφισμα που αναφερόταν στην τάση αυτή, στον χειρισμό αυτό και λέγαμε ότι ναι, μεν εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εμείς το είχαμε πει ξεκάθαρα ότι προσοχή. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ, δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στα τυφλά, πρέπει να καθίσουμε να εξετάσουμε πάρα πολύ καλά τι επιπτώσεις μπορεί να έχει ένα τέτοιος μηχανισμός και θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι εμπλεκόμενο. Τι είπε δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε ότι όσον αφορά τους στόχους, πέρα από την μείωση της ένδυας και την καταπολέμηση των αδικιών, το κράτος πρέπει να είναι σε κεντρικό σημείο. Θέλουμε λοιπόν φτώχεια, καταπολέμηση της φτώχειας, καταπολέμηση ανισοτήτων και τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται με το συνδυασμό αυτό να σέβονται τους αναπτυξιακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρεται στους αναπτυξιακούς μας στόχους δηλαδή. Έχουμε πει και το τονίζω ότι πρέπει να ελέγχει το Κοινοβούλιο το τι γίνεται. Μετά περάσαμε στην πλατφόρμα αυτή που μας εξήγησε τώρα ο κύριος Μοραθών και τον ευχαριστώ για την μελέτη. Είναι εξής το κόπο, το διαβάσετε, δεν είναι και τόσο μεγάλο με 40 σελίδες, διαβάζετε εδώ ολόκληρη την προβληματική και διαβάζετε ευχάριστα το κείμενο. Έγινε μία πολιτική συνάντηση στην αρχή, μετά υπάρχουν οι τεχνικές συναντήσεις, τις οποίες εκπροσωπούμε εμείς από την γραμματεία της Επιτροπής μας. Η επόμενη συνάντηση είναι στις 21 Ιουνίου, η πολιτική. Και εδώ έχω κάποιες ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα, ναι, έχω έξι. Πρώτον, όσον αφορά την διακυβέρνηση, την ε, διαχείριση δηλαδή του μηχανισμού αυτού. Γιατί διαπιστώσαμε ότι λιγότερο από 50% των περιπτώσεων εντοπίζονται ως να, ένα πρόγραμμα, από τα προγράμματα τα οποία μάλλον μπορούν να είναι για συνδυασμό, συμμετέχουν πολύ λίγες αντιπροσωπείες. Δεν εντοπίζουν δηλαδή οι αντιπροσωπείες τα προγράμματα. Κινδυνεύουν δηλαδή να πρόκειται για τεράστια προγράμματα Σήμερα το πρωί μίλησα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη λέει Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση, υπάρχει μια εξέλιξη με τα χρόνια, βελτιώνεται η κατάσταση. Αλλά λέει ότι πρέπει οι αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν πιο δραστήρια, να εμπλέκονται περισσότερο. Υπάρχει ο του προγράμματος, αλλά δεν μπορεί να εντοπίζεται ένα πρόγραμμα για συνδυασμένη χρηματοδότηση χωρίς να εμπλέκεται η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερον, εμπλοκή του ντόπιου πληθυσμού. Είτε πρόκειται για τον ιδιωτικό, είτε για το δημόσιο τομέα, είτε πρόκειται για την κοινωνία των πολιτών, πρέπει να εμπλέκονται και αυτοί. Εμεί το θέλαμε αυτό. Είναι βασικό στόχο τη αναπτυξιακή μα πολιτική Υπάρχει και στη Λισαβόνα κλπ. Οι τοπικοί φορεί, λοιπόν, πρέπει να εμπλέκονται και να συμμετέχουν, ενώ από ό,τι φαίνεται δεν συμμετέχουν και δεν εμπλέκονται συστηματικά για τον καθορισμό των προγραμμάτων. Τρίτον, τρίτο πρόβλημα. Εμείς είπαμε, και το λέει και η μελέτη, το είπατε κι εσείς, πρόκειται για τις μελέτες επιπτώσεων εξάντε όσον αφορά την άδεια, που πρέπει να γίνονται συστηματικά βάσει κριτηρίων. Ο καθένας να μπορεί να τα διαβάσει και να τα καταλάβει και να μπορεί να πάρει κάποια στοιχεία από την αξιολόγηση αυτή που θα γίνεται βάσει κριτηρίων. Επόμενο, δεν είναι σαφές ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε κάποια σύσταση. Τέταρτη ανησυχία μου. Οικονομική πτυχή. Υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οργανισμοί που χρηματοδοτούν με, το με τη συνδυασμένη χρηματοδότηση θα ακολουθήσουν τις τάσεις που επικρατούν στον οικονομικό τομέα, δηλαδή τις τάσεις της αγοράς. Οπότε θα επικεντρωθούν στην οικονομική ανάπτυξη. Και σε μηχανισμούς οι οποίοι αποδίδουν περισσότερο, που χρησιμοποιούν συνήθως ε, όλοι στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό είναι ο φόβος μου, ότι αν μπούμε σε αυτή τη λογική, τότε στο τέλος δεν θα υπάρχει ισορροπία, δεν θα υπάρχει μια ανάπτυξη για όλους και οι επιπτώσεις υπέρ της απάλληψης της φτώχειας δεν θα είναι ίδιες. Στο μηχανισμό αυτό δηλαδή συνδυασμένης ε, χρηματοδότησης δεν δίνεται η προσοχή που θα έπρεπε στις μικρές επιχειρήσεις, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στις υποδομές, στην ενέργεια κλπ. κλπ. Πέμπτη ανησυχία μου. Είδαμε ότι στις συζητήσεις που γίνονται στην πλατφόρμα δίνουμε λίγη προσοχή στις επιπτώσεις πραγματικά υπέρ της απάλληψης της στόχιας. Εδώ πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να καθοριστούν δείκτες οι οποίοι να φροντίζουν που να έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της ένδυας, έτσι, και οι οποίοι δείκτες να χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση. Έκτη και τελευταία μου ανησυχία. Είναι σαφές ότι η συνοχή ε, δεν είναι πάντα παρούσα της πολιτικής μας. Έχουμε πολλοί τομεί. Ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, υπάρχει Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνέ Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν διαφορετικά οράματα, διαφορετικέ απόψει. Από πλευρά τη Κομισιόν και τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσει, αν μη τι άλλο, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει συνοχή όσον αφορά την πολιτική μα για την συνδυασμένη χρηματοδότηση. Συνεπώ, εν κατακλείδη, η ανησυχία που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο ότι η καταπολέμηση της ένδυας είναι πραγματικά ο κατεξοχήν στόχος της συνδυασμένης χρηματοδότησης. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει παραπάνω δουλειά, αξιολόγηση του τι γίνεται. Και, και αυτή είναι μια κριτική μου επίσης, ότι δεν συμμετέχει αρκετά η κοινωνία των πολιτών αυτό λείπει. Η όλη διαδικασία λαμβάνει η χώρα μέσα σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Υπάρχουν βέβαια οι ευρωβουλευτές που μπορούν να είναι παρατηρητές, αλλά αυτό για μένα είναι προβληματικό. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων, τα συμπεράσματά τους πρέπει να είναι κατανοητά για όλους. Και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα συμπεράσματα της πλατφόρμας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα είμαστε παρατηρητές, λίγο μπορεί να επηρεάσει. Ακούω ότι εκτός από το Βέλγιο οι περισσότερες χώρες δεν συμμετέχουν καν. Σας είπα, δεν υπάρχει παρουσία της, Επιτροπή, της Κοινωνίας των Πολιτών. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Πίβελξ. Και έχω μια έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών πρέπει να θέσουμε κάποια ερωτήματα στον κύριο Πίβικαλης. Θα υπάρξει ανακοίνωση της Επιτροπής για αυτό το θέμα. Πώς θα συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του Οκτωβρίου. Πρέπει να ρωτήσουμε λοιπόν τον κύριο Πίμπαγκ για όλες αυτές τις ανησυχίες, τις δικές μου αλλά και των συναδέρφων που φαντάζομαι θα ακουστούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κόρτες Λάστρα, έχετε στήσει το λόγο. Ε, σύντομο πρόεδρε, διότι παρευρίσκεται και η Επίτροπος παρούσα, να ευχαριστήσω τον κύριο Μοναθάν για την έκθεση, αλλά και τον κύριο Στάις. Νομίζω ότι έκαναν παρεμβάσει πληρέστατες, αλλά έχουμε την εντύπωση τουλάχιστον ορισμένη εξίμων βρισκόμαστε ενώπιον μιας ευκαιρία που όμως ε, συγχρόνως αποτελεί και ε, ένα μεγάλο κίνδυνο. Ο τρόπος με τον οποίο θα δουλέψουμε σε ό,τι αφορά το συνδυασμό των επιχορηγήσεων για δανείο και τη χρηματοδότηση μπορούμε μια φορά να περάσουμε και στο θέμα της ε, διεθνούς βοήθειας, το κώδικα συμπεριφοράς που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για όλες αυτές τις ιδιωτικές επενδύσεις που αφορούν τον τομέα της ανάπτυξης και είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός. Έχουμε ένα συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς και δεν μπορούν να ρυθμιστούν με έναν γενικό Δεν Θέλω να τονίζω αυτό το σημείο, διότι η συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Στον τομέα της συνεργασίας μιλάμε πολύ για οικονομική και δημόσια συνεργασία, εμπλέκεται και θέματα, θέματα ασφαλείας κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια αναδιάταξη της έννοιας ε, της συνεργασίας και της ε, βοήθειας που δίνεται. Πρέπει να είμαστε λοιπόν, λοιπόν πολύ προσεκτικοί ώστε να μην ε, βρεθούμε ενώπιον εκπλήξεων. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο για λίγο χρόνο. έχω καθυστερήσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο κύριος Καράνο για δύο λεπτά και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Μπέκ για άλλα δύο λεπτά. Κύριε Καράνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω ε, αυτούς που έγραψαν τη μελέτη και τον κύριο Στάση για τις παρατηρήσεις του συμμετέχουμε ενεργά στην πλατφόρμα και πλησιάζουμε σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τον καθορισμό κάποιων παραμέτρων για τον καθορισμό του αντικτύπου των προγραμμάτων και έχει δημιουργηθεί ειδική υποομάδα υπό την πλατφόρμα και συνεργαζόμαστε και με τα άλλα θεσμικά όργανα η Κομισιόν προεδρεύει στις εργασίες για να βελτιωθούν ε, τα διάφορα στοιχεία των ε, συστημάτων συνδυασμού. Γενικά, στηρίζουμε τον συνδυασμό εφόσον συνδέεται με τους πολιτικούς στόχους και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η βασική ανησυχία μας. Επίση, μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να διασφαλίσουμε την ορατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός ε, συνδυασμού μπορεί να δώσει περισσότερη ορατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν συμμετέχουμε σε ε, προγράμματα ε, χρηματοδοτικά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μπορέσουμε να δείξουμε ε, τον αντίκτυπο των προγραμμάτων αυτών. Αυτό θα είναι δυνατό όσο θα συλλέγουμε περισσότερα ε, δεδομένα ε, χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Και επίσης πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα περισσότερης μόχλευσης και οικονομικής και πολιτικής. Με την πείρα μας έχουμε διαπιστώσει ότι μπορούμε να προσελκύσουμε χρηματοδότηση όχι μόνο από άλλους οικονομικούς οργανισμούς αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα και από ιδιωτικά ιδρύματα και πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα μόχλευσης όσον αφορά την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν τα χρησιμοποιήσουμε αυτά στους διαλόγους μας με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κομισιόν, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανάπτυξης που μας προσκάλεσε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρθέν για την ε, μελέτη του. Συμμεριζόμαστε τα περισσότερα επιχειρήματά του. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Στάς και τον κύριο Κορτές για τις παρατηρήσεις τους. Είχα ετοιμάσει μια ε, ε, κάπως πιο μακρά παρέμβαση, αλλά θα περιοριστώ στα απαραίτητα. Καταρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω ή να τονίσω ότι ο μηχανισμός συνδυασμού πάντα βρίσκεται εντός των πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διασφαλίζουμε. Οι τομείς στους οποίους εργαζόμαστε, ενέργεια, μεταφορές, ε, υποδομές, ε, ο κοινωνικός τομέας ενδεχομένως, είναι τομείς που ε, έχουν ε, εντοπιστεί ως ε, επιλέξιμοι και συμβάλλουν στην μείωση της φτώχειας. Κάνουμε σοβαρή δουλειά στο πλαίσιο της πλατφόρμας. Προσπαθούμε να εκπονήσουμε δείκτες που μας επιτρέψουν να εξετάσουμε τον αντίκτυπο των προγραμμάτων. Έχουμε καταλήξει σε κάποια συμφωνία με, τους, με χρηματοπιστωτικό οργανισμό σχετικά με του δείκτε αυτού και θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ε, ένα βήμα πιο πέρα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Έχει γίνει πολλή συζήτηση σχετικά με την χρήση δικτών ε, ε, όσον αφορά τα άλλα στοιχεία συνεργασία, αλλά τελικά δεν έχουμε καταλήξει σε κάτι οριστικό, αλλά οδεύουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να τονίσω ότι μία οδηγία μας ε, προς ε, τους ε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς είναι ότι θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις αντιπροσωπείες μας ήδη από την αρχή των προγραμμάτων ώστε να διασφαλίζουμε, να διασφαλίσουμε την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών στα προγράμματα αυτά. Πιστεύω ότι οι μηχανισμοί συνδυασμού μας δίνουν μια εξαιρετική ευκαιρία συντονισμού των προσπαθειών ε, διαφόρων παραγόντων, όχι μόνο των χρηματοπιστωτικών ε, οργανισμών, αλλά και άλλων οργανισμών. Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να απορρίψουμε τη δυνατότητα αυτή στο μέλλον. Τέλος. Ε, έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Επιτρέψτε μου να πω ότι οι μηχανισμοί συνδυασμού ε, και μόνο λόγω του γεγονότος ότι έχουν να κάνουν με την υποδομή επιτρέπουν ε, να δοθεί περισσότερη ορατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. τον κύριο που ήρθε ανάμεσά μας και τον κύριο που πρόθεσε τις ανησυχίες ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πλατφόρμας και μετέφερε τις θέσεις μας και τέλος προς την Κομισιόν να πω ότι καλό θα ήταν να συντάξετε επί του ζητήματος του συνδυασμού επιχορηγήσεων μια έκθεση προκειμένου να επιτρέψετε στο Ευρωκοινοβούλιο να αντιδράσει επισήμως. Και τώρα θα μιλήσουμε για τον διαφρομένο διάλογο σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014. Πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό στην μεσαιριάταξή διάταξή μας να γνωρίζουμε το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2014 σε ό,τι αφορά ανθρωπιστική βοήθεια και για τον λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας την Επίτροπο κυρία Κρυσταλίνα Γεώργιεβα. Θα ενθυμίστε πως η συμφωνία πλαίσιο που έχει υπογραφεί από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν τον Οκτώβριο 2010 επιτρέπει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές να υποδεικνύουν τις δραστηριότητες που θα ήθελε να αναλυφθούν από πλευράς Κομισιόν κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς. Έχουμε κληθεί φέτος να συζητήσουμε το πρόγραμμα της Κομισιόν για το 2014 αλλά και να αξιολογήσουμε την νομοθεσία και τις δεσμεύσεις που έχει λάβει η Κομισιόν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περίοδου για να δούμε κατά πώς να τα αποκρίνονται στις προτεραιότητες της Επιτροπής μας και που δεν απουσιάζουν κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίε. Επίσης αναφέρεται ότι οι νομοθετικές διαδικασίες και ιδίως οι πιο σημαντικοί για μας που αφορά την ε, Κομισιόν. Αύριο θα έχουμε τον ε, διάλογο με τον κύριο Σπίμπαλς, τον Επίτροπο, και μετά από τις συζητήσεις αυτές με τους δύο επιτρόπους, οι συντονιστές μας θα αποφασίσουν τις ε, συστάσεις που θα στείλουν στους διάσκεψεις των Προέδρων των Επιτροπών σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014. Κυρία Επίτροπε, ε, θα μας παρουσιάσετε αρχικά τις προτάσεις της Κομισιόν και τις ιδέες σας ε, για το 2014 και μετά θα μπορέσετε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή αυτού του πρόγραμματος κατά το 2013 αλλά και κατά τις προηγούμενες χρονιές. Επίσης μπορείτε να κάνετε ε, προτάσεις για την πρόγραμμα της προσεχούς χρονιάς. Να συμπεριθυμίσω ότι η σημερινή ανταλλαγή απόψεων δεν είναι μια τακτική ανταλλαγή απόψεων επί του ανθρωπιστικού προγράμματος ή την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων σε ε, περιοχές του κόσμου. Η συζήτηση μας θα πρέπει να εστιαστεί αποκλειστικά στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν. Κυρία Γιορτζεβα, σας δίνω το λόγο. Ε, merci, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, πάντα όταν έρχομαι στην Επιτροπή σας ε, ε, γνωρίζω πως θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και επιτρέψτε μου να διαδρώσω την παρέμβασή μου σε τρία σημεία. Πρώτον, πώς θα αντιμετωπίζουμε τα κατεπίγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ε, ανάγκες. Ε, δεύτερον, πώς προωθούμε τη ε, νομοθετική μας ατζέντα. Πολλά πρέπει, έχουν να γίνουν φέτος. Το 2014 θα δούμε και τους καρπούς αυτής της νομοθεσίας. Επίσης, ό,τι φορά τις πολιτικές, τις πολιτικές προτεραιότητες για το 2014, αλλά και τρίτον, τι κάνουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ε, οι δεσμεύσει μας ε, σε ό,τι αφορά στους εθνικού προπολογισμού θα προσφέρουν το δυνατό μεγαλύτερη προσθέμενη αξία για την ανθρωπιστική βοήθεια και για την διεθνή συνεργασία. Δηλαδή πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τη δράση μας και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα από τα 2014 τώρα σε ό,τι φορά το θέμα της, ε, των ανθρωπιστικών προτεραιοτήτων φέτος, του χρόνου και τα επόμενα χρόνια αυτό το ζήτημα νομίζω θα πρέπει να παραμείνει υπαριθμόν ένα προτεραιότητα. Πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τους περισσότερους δυνατούς ανθρώπους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές με τον, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Να σας δώσω κάποια δείγματα της πρόοδου που πετύχαμε, μια πρόοδος η οποία φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον με τον επόμενο Επίτροπο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Καταρχήν, προβλέπουμε στις αρχές του έτους για τις κρίσεις τις οποίες γνωρίζουμε πόρους που θα δώσουμε στις αποφάσεις που έχει λάβει το Κοινοβούλιο και σας είμαι ευγνώμονος για τη συμμετοχή σας. Αυτό θα μας επιτρέψει τρία τέταρτα ή να τα δύο τρίτα του προπολογισμού στις αρχές Ιανουαρίου και να προσδιορίσουμε τις προτεραιότητες τις οποίες γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανάγκες ήδη. Το πράξαμε πέρυσι, φέτος τα πράγματα πήγαν καλύτερα διότι ορίμασαν και ελπίζουμε του χρόνου η διαδικασία θα ολοκληρωθεί και θα μπορούμε να προβλέψουμε και τις μελλοντικές ανθρωπιστικές ανάγκες με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούμε τους εταίρους να μπορούν να έχουν δυνατότητα πρόληψης και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από αυτή τη βοήθεια και ότι θα είμαστε παρόντες. Φέτος στην απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότηση έχουμε το Σουδάν, την Σομαλία, το Αφγανιστάν, μόνο για να αναφέρω μερικά από τα κράτη, και το, ίδιο θα συμβεί και την επόμενη χρονιά. Μακάρι να μπορούσα να είχα κάνει μια διαφορετική πρόληψη. Το μόνο πράγμα που θα αλλάξει είναι ότι αυτά τα οποία θα γνωρίζουμε στι αρχέ του επόμενου έτου, αναφορικά με τι κρίσει αυτέ που δυστυχώ παρατείνονται και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, ε, συνεργάτες μου και από τον πρόεδρο Μπαρόζο ότι η βοήθεια που λάβαμε για την καταπολέμηση αυτών των κρίσεων δεν, ε, δεν παραμελούνται, δεν ξεχνιούνται, θα συνεχίσουμε του χρόνου όπως το πράξαμε και φέτος ε, και να, για να είμαστε βέβαιοι όταν προκύπτουν κάποιες ε, δραματικές κρίσεις εμείς στην Ευρώπη θα μπορούμε να διαρμονίσουμε έναν τριπλό ρόλο της στήριξης, ε, της ε, εποπτείας ε, και της παροχής βοήθειας. Φέτος ήταν η Συρία, το Μαλί, Κεντρική Αφρική, που μας οδήγησαν στην πρώτη θέση σε φορά την βοήθεια που παρέχει η Ευρώπη σε αυτές τις κράτη και Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω ότι κάναμε πολλά πράγματα, διότι δυστυχώς η κρίση στην Συρία ε, μεγεθύνεται όλο και περισσότερο, περισσότερο από τις ικανότητες που έχουμε. Αν ε, κάποιος έχει προχωρήσει, αυτή είναι η Ευρώπη. 865 εκατομμύρια ευρώ, 65 εκατομμύρια τα ανήγγυλα που τα εβδομάδες για την Ιορδανία και το Λίβανο και είμαστε ε, ένα περιοχή που δρά ε, στις χώρες αυτές. Φοβούμε όμως ότι και του χρόνου θα χρειαστεί να δουλεύουμε πάνω σε αυτές τις, αυτά τα δύο κράτη. Τώρα έχουμε 500 περίπου 5 εκατομμύρια άτομα που έχουν ε, μετακινηθεί στο εσωτερικό. 700.000 ε, πρόσφυγες ε, στην Συρία και 2 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Η κατάσταση είναι πιο τραγική ακόμα και αυτή που υπήρχε στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία και η κρίση πραγματικά έχει αρχίσει να επεκτείνεται στην περιοχή αυτή της Μέση Ανατολής. Στο Μαλί φέτος ε, δράσαμε αποτελεσματικά 125 εκατομμύρια ε, ευρώ χορηγήσαμε. Κοιτάζοντα όμω ε, την κατάσταση τη περιοχή αυτή, βλέπουμε ότι εδώ θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προτεραιότητα. Το ευάλωτο αυτών των περιοχών και το έφραστο χαρακτήρα δείχνει ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ε, διατροφή των παιδιών θα επιδεινωθεί. Τώρα σε ό,τι αφορά το δεύτερο κομμάτι του προγραμματός μας, ε, νομοθετικές προτάσεις. Ε, έχουμε δύο νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ελπίζουμε πως θα τις ολοκληρώσουμε το 2013 και θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή τους το 2014. Πρώτα αυτά ό,τι αφορά την νομοθεσία για την πολιτική προστασία κάναμε σημαντικές προόδους και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στρίφτερ αλλά και την Επιτροπή σας στο σύνολό για την υποστήριξη της οποίας είχαμε και επειδή του περιβάλλοντος ήταν ιδιαίτερα ενεργή όπως και εσείς. το κέντρο αντιμετώπισης ε, των ε, εκτάσεων καταστάσεων δείχνει ότι βελτιώνουμε τις δυνατότητές μας ε, να ανταποκριθούμε σε έκτακτες καταστάσεις και θα θέλω να καλέσω την κυρία Ζωλή να έρθει και να επισκεφθεί όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής το κέντρο για να δείτε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανθρωπιστικές κρίσεις και σε άλλες καταστροφές. Δεύτερη νομοθετική πρόταση είναι η UAID Volunteers, οι εθελοντές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ η κυρία Στίφταρ ήταν ιδιαίτερα ε, επικοδομητική στη δράση της αντιμετωπίζουμε μια πολύ σκληρή κατάσταση διότι ο προπλοισμός έχει τύχει περικοπών, κάναμε επιλογές και κάναμε επιλογές υπέρ της προστασίας του επιχειρησιακού προϋπολογισμού μας. Αυτό σημαίνει ότι το περιφερειακό φάκελος είναι τώρα μικρότερο πιο περιορισμένο. αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή νομοθεσία που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει πλατφόρμα για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας μόλον ότι ακόμα δεν έχουμε αναπτύξει ταχύτητα. Ελπίζω πως στα τέλη της χρονιάς θα έχουμε πετύχει την απαραίτητη πρόοδο και του χρόνου θα περάσουμε στην εφαρμογή. Το μισό όπου θα δείτε το 2014 να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά ψήφα της πολιτικής πρωτοβουλίας είναι τέσσερις. Πρώτον, θα προωθήσουμε την συνεργασία για το πώς ε, μπορούμε να καταστήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια κατάλληλη για το στόχο για τον 21ο ε, αιώνα. Έχουμε περισσότερους προορισμούς από πλευρά πόρων και αυτό τα οποία κάνουμε θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη ε, να υποφελούν ιδιαίτερα από τα κονδύλια τα οποία παρέχουμε και να μην γίνονται σπατάλες. Ε, τώρα τον Ιούνιο θα έχουν μια διαδικασία προκειμένου να προετοιμάσουμε και τον διάσκεψη κορυφή του 2015 για την ανθρωπιστική διάσκεψη. Δεύτερον είναι το ζήτημα της ε, ατζέντα ε, που έχει θέσει ο κύριος Σπίλμπαρκ Spielberg εργαζόμαστε με ένα πρόγραμμα δράσης και αυτό που θέλουμε 2014 είναι να δούμε μια καλύτερη εφαρμογή στα δύο σημαντικά προγράμματα που έχουμε προωθήσει για την περιοχή του Σαχέλ και για το γέρα της Αφρικής αλλά και πρόοδο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δράσης για τις χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτε όπως IT, εμένη κλπ. Τρίτον, ζητήθηκε από την Επιτροπή σας να συνεργαστούμε πάνω σε θέματα ε, ανάπτυξης και αποκατάστασης Το 2014 αυτό το οποίο θα προχωρήσει είναι η βελτίωση της χρηματοδότησης στα κράτη που είναι πιο ευάλωτα για ε, ε, ε, συγκρούσεις, εθνοτικές συγκρούσεις. Τέλος, αλλά λιγότερο σημαντικό, οι διάφορε ε, πολιτικές που έχουμε, πρωτοβουλίες, που έχουμε αναλάβει για τις πιο ευάλωτε ομάδες όπω γυναίκε, παιδιά και πληθυσμού που έχουν πληγεί από υποσυτισμό. Ο Επίτροπος Πίλμπαρξ ε, έχει κάνει νέες ανακοινώσεις σε αυτούς τους τομείς ε, και τώρα θέλουμε να μετατρέψω αυτές τις ανακοινώσεις σε ε, δράσεις να εστιαστούμε περισσότερο στα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. σε συγκεκριμένα προγράμματα στις χώρες όπου συμμετέχουμε σε παροχή ανθρωπικής βοήθειας. Γνωρίζετε πως εξετάσαμε κατά πόσο θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν βρήκαμε πιστικούς λόγους προκειμένου να το πράξουμε Δεν κρίνουμε λοιπόν που θα έπρεπε να διορθώσουμε κάτι το οποίο δεν έχει σπάσει, δεν έχει ραγίσει. Ξεκινήσαμε μια διαβούλευση, δεν την έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Θα την ολοκληρώσουμε στα τέλη Ιουνίου. Δεν θέλω να προκαταλάβω τα τελικά αποτελέσματα, αλλά μέχρι τώρα στη διαδικασία διαβούλευσης δεν υπήρξαν αξιόπιστες ενδείξεις ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τον κανονισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Τέλος, τι κάνουμε για να βεβαιωθούμε ότι δεν ζητάμε από τους άλλους να είναι αποτελεσματικοί μόνο, αλλά και από τους εαυτούς μας Είχαμε την ε, διαδικασία εξέτασης προόδου και προερθέμεθα να πετύχουμε μια αύξηση της, ε, των επιδόσεων μας κατά 15-20% τα επόμενα πέντε χρόνια. Να κάνουμε λοιπόν ε, περισσότερα και καλύτερα με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας ξεκινήσαμε ε, την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. Ε, η επόμενη χρονιά θα είναι κρίσιμη για την εφαρμογή. Πολλοί από τους συνάδελφους μου ε, ανησυχούν πως αυτή η διαδικασία θα αποτελέσει την μητέρα των όλων διαδικασιών, αλλά θα πρέπει οι υπηρεσίες μου να ζητήσουν από τους εταίρους μας να συνεργαστούν προκειμένου να καταστούν και αυτοί αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι. Πώς λοιπόν μπορούμε να δράσουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα μέσα στο πλαίσιο των περιορισμένων πόρων επαναλαμβάνω που έχουμε στη διάθεσή μας. και να τελειώσω λέγοντας πως ε, τα τελευταία χρόνια ε, έγιναν διάφορες θεσμικές αλλαγές λόγω της δημιουργίας της, εξωτερικής, της υπηρεσίας μάλλον δράσης και λόγω της μείωσης των πόρων. Μια καλή πρόοδος όμως επιτεύχθη συνεργαστήκαμε στενά με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και επίσης με τους συναδέλφους στον τομέα της ανάπτυξης. Κοιτάζοντας λοιπόν λίγο πίσω, μια από του χρόνου λίγη θητεία μου και θα είναι κρίσιμη χρονιά, θα αφήσουμε μια υπηρεσία πολιτικής προστασίας ικανοποιητική πολλά οφείλονται στους συναδέλφους μου στην ΕΚΟ μεταξύ των πολύπτων προσωπείων που βρίσκονται στην αίθουσα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το έργο σας. Είναι ένα έργο το οποίο φέρεται σε πέρασμα όλο και λιγότερους σπόρους. Οπότε βέβαια είναι πολύ δύσκολο να κατηγορήσει κανείς την ε, Ευρώπη όταν πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια. Βέβαια, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια βοήθεια αμερόληπτη, ανεξάρτηση και από μόνες τους οι χώρες μέλη δεν θα καταφέραν να φτάνει η βοήθειά του στον προορισμό της. Και αυτό είναι προστιθέμενη αξία. Η ανθρωπιστική βοήθεια πάντως, που όλοι συμφωνούμε με αυτήν, είναι κάτι που δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Δεν μπορεί δηλαδή να μειώνεται ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πάει σε ανθρωπιστική βοήθεια. Με τίποτα. Εγώ είμαι από αυτού που πιστεύουν ότι στι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ και ένα ευρώ να μειωθεί σε ανθρωπιστική βοήθεια θα έπρεπε να καταψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις δημοσιονομικές προοπτικές. Γιατί έχει να κάνει και με το πνεύμα, με τις αξίες, με το τι είναι στην ουσία η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πιστεύω, 550 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. είναι πάρα πολλοί κόσμος σε ολόκληρο το κόσμο και αυτά τα παιδιά στα οποία αναφερθήκατε κάτω το 5 ετών. Και αυτούς θέλουμε να στηρίξουμε, παιδιά, γυναίκες και άλλες ευάλωτες ομάδες που έχουν περισσότερες ανάγκες. Έχουμε και ηθικό χρέος να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά είναι και μια υποχρέωση που έχουμε αναλάβει απέναντι στην κοινωνία μας, που ξεπερνάει βέβαια τα σύνορά μας. Για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν στον κόσμο. Έχουμε πολλούς στόχους μπροστά μας. Υπάρχει ο διαρθρωμένος ο διάλογος, αλλά αυτό ίσως να είναι το πιο δύσκολο, το πιο περίπλοκο θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί του χρόνου. Μπορεί να έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα. Πάντως την ευελιξία τη χρειαζόμαστε αυτή στην οποία αναφερθήκατε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και τα νέα που θα μας προκύψουν είναι μια συζήτηση που ίσως θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο σε βάθος εδώ. Δεν είναι δυνατόν σήμερα η ανθρωπιστική βοήθεια να μειωθεί στις δημοσιονομικές προοπτικές. Δεν γίνεται. Το πιστεύω πραγματικά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Τι θα γίνει στη συνέχεια. Ήδη κανένας δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι τα ποσά. Άρα υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα για τα ποσά. Πάντως, αν υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο να αγωνιστούμε γι' αυτό, είναι η ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, μας την εξηγήσατε και για την οποία νιώθουμε όλοι περήφανοι και που βασίζεται στις αξίες και στην ουσία την ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι πάντα δύσκολο να παίρνει κανείς το λόγο μετά από την κυρία Γιώργεβα, διότι είναι πάντα πλήρης σε αυτά που μας λέει. Πολλοί από μας στην Ολομέλεια στηρίξαμε τη θέση σας όταν μιλούσαμε για τη Συρία. Μια κατάσταση φρικτή. Αλλά ξέρω ότι η υπηρεσία σας κάνει ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί με τα μέσα βέβαια που έχετε στη διάθεσή σας. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, η συμπληρωματικότητα ανάμεσα στη δικιά σας δράση και εκείνη των κρατών μελών. Δεν πιστεύετε πως ήρθε ο χρόνος, ο καιρός, να κάνουμε μια αξιολόγηση για την ανάγκη της συμπληρωματικότητας αυτής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Πήγα στην Επιτροπή προπολογισμών για να ζητήσω από τον κύριο Λαμασούρ να ετοιμάσει την επιστολή της κυρίας Ζολή και την Κυρπό για την συνεισφορά των κρατών μελών. Δεδομένου ότι οι πόροι που έχετε εσείς στη διάθεσή σας εξαντλούνται. Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και να συμπληρώσουν 28 όλοι μαζί τις ανάγκες που υπάρχουν. Δεύτερον, διπλωματική δράση από κοινού με άλλους. Τι κάνουν οι αραβικές χώρες. Κάνουν κάτι πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι κάνουν αρκετά. Η θέση που εσείς ως Επίτροπος έχετε στα διεθνή φόρα και που ανταποκρίνονται στην ανάγκη για αμεροληψία, μπορείτε να πείσετε και άλλους. Νιώθετε λοιπόν ότι οι συναδελφοί σας και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης που σας στηρίζουν αρκετά για να προσπαθήσετε να πείσετε και τους άλλους. Ή από ποια στιγμή η στήριξη των άλλων, δεδομένου ότι εσείς είσαστε υπέρ της αμεροληψίας, η στήριξη αυτή μπορεί να σας δυσκολέψει στο στόχο αυτό. Τρίτον, Υπογραμμίζω και πάλι ότι πρέπει η αρχή της αμεροληψίας να τηρηθεί πλήρως και απόλυτα. Ξέρουμε τα νέα, τα παρακολουθούμε, δεν υπάρχουν πια λόγια να περιγράψει κανείς την κατάσταση. Παρακολουθούμε και προσπαθούμε με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας να φροντίσουμε να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να βάλουν το πετραδάκι τους για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βασίλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Φυσικά όπως είπε ο κύριο Γκέρεν, είναι, να πάρει, είναι δύσκολο να πάρει κανεί το λόγο μετά από εσά, ε, αλλά είναι ακόμη πιο δύσκολο να μιλήσει μετά από αυτόν, διότι αυτός κάλυψε τα περισσότερα θέματα που ήθελα να θίξω και εγώ, αλλά θα ήθελα να διευρύνω την ερώτηση του κυρίου Γκέρενς σχετικά με την αλληλεγγύη εργασία. Ήθελα να ρωτήσω, η κρίση είναι σε αυξανόμενο βαθμό παγκόσμια. Και βλέπουμε να γίνεται όλο και περισσότερο παγκόσμιο πρόβλημα οι καταστροφές. Θα έχουμε περισσότερες στο μέλλον. Έχουμε παγκόσμια αλληλεγγύη και παγκόσμια συνεργασία. Και δεν μιλώ μόνο ε, για τις χώρες του κόρπου, μιλάω για τις χώρες BRICS, έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες, έχουμε... Πολλές χώρες που σίγουρα θα έπρεπε να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μοιράζονται το βάρος της αλληλεγγύης. Σίγουρα είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεχίζει να ηγείται στο χώρο ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας και βέβαια ε, ε, η επιτυχία αυτή οφείλεται και σε εσά, ε, στο γραφείο σας και σε εσά προσωπικά και θα ήθελα να σας επενέσω γι' αυτό. Από την άλλη όμως έχουμε ένα πολύ έντονο πρόβλημα με τη Συρία. Στη Συρία δεν έχουμε φυσική καταστροφή, έχουμε μια καταστροφή που οφείλεται στον άνθρωπο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτική οντότητα δεν έχει ε, να δείξει αποτελέσματα. Ε, τώρα έχουμε τη διεθνή διάσκεψη που θα προσπαθήσει να βρει πολιτική λύση, αλλά η πολιτική αυτή λύση θα ήταν δυνατό να είχε επιτευχθεί πριν δύο χρόνια, διότι ήταν ε, ήδη τότε σαφές προς ποια κατεύθυνση θα πηγαίναν τα πράγματα. Πρόσφατα, εδώ στο Κοινοβούλιο, είχαμε συζήτηση με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Και εγώ του έθεσα μία ερώτηση, την οποία εκείνος δεν απάντησε. Προσπαθούσε να μας πείσει ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα πρέπει να εκφράζεται ως περισσότερες δαπάνες για όπλα και μοίρασμα των ε, δαπανών στον τομέα αυτών. Και εγώ τον ρώτησα, ε, και τι γίνεται με την αλληλεγγύη που εκφράζεται όχι ε, σε περισσότερα χρήματα, αλλά περισσότερη σοφία, περισσότερη ευφυΐα και δυνατότητα να προβλέψει κανείς τις νέες καταστάσεις, διότι αυτός είπε ότι καθήκον μας είναι να είμαστε έτοιμοι ε, και σε περίπτωση απροσδόκητων κρίσεων και γεγονότων. Και του είπα ναι, αλλά ξέρετε, Αντί να έχουμε λιγότερα προσδόκητα γεγονότα, έχουμε περισσότερα. Και δεν χρησιμοποιούμε τις δυνατότητές μας για να προβλέψουμε τις κρίσεις και τα προβλήματα. Και δεν προσπαθώ τώρα να μαντέψω που θα προκύψει η επόμενη ε, πολιτική κρίση που μετά θα γίνει στρατιωτική και ανθρωπιστική. Αλλά ξέρουμε λίγο πολύ που υπάρχουν κρίσεις, που υπάρχουν ε, ε, παγωμένες διαμάχες, να το πούμε έτσι, και κάνουμε πολύ λίγα πράγματα για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Ε, μπορεί να έχουμε αυτές τις λεγόμενες παγωμένες διαμάχες, ε, ξαφνικά όμως ε, μπορεί να θερμαίνεται η κατάσταση. Και κύριε Επίτροπε, Ε, μπορεί να μην είναι μια συζήτηση που πρέπει να διεξάγουμε μαζί σας, αλλά εσείς εμφανίζεστε στο τέλος του προβλήματος για να πληρώσετε το λογαριασμό, όπως όλοι μας. Για το λόγο ότι δεν ήμασταν αρκετά προορατικοί και προληπτικοί. Ελπίζω Ε, να μπορείτε να αντιληφθείτε τις ε, σκέψεις μου ως ερώτηση προς εσάς και να τις σχολιάσετε. Ευχαριστούμε, η ε, κυρία Γκρέση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που άργησα, αλλά ήμουνα σε μια άλλη επιτροπή όπου πήρα το λόγο. Θέλω να επανέλθω στο θέμα των προσφύγων εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές και οι καταστροφές αυτές αυξάνονται. Κύριε Γεώργιεβα, θυμάμαι ότι όταν ήσασταν στην Παγκόσμια Τράπεζα σε κάποια παρέμβασή σας είχατε πει ότι στηρίζετε τον αγώνα που γίνεται κατά της αποψήλωσης των δασών. Ως επίτροπος τώρα, από τη θέση αυτή, τι έχετε κάνει όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Τι κάνατε για να αποφύγουμε τέτοιους πρόσφυγες εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Και θέλω επίσης την αναλυσή σας, την άποψή σας και πώς απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόβλημα αυτό των προσφύγων εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Γεώργιεβα, θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι. Για τη Συρία. Γνωρίζουμε ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Ξέρουμε επίσης ότι πριν από τα τέλη της χρονιάς θα έχουμε 3,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα οργάνωσης είναι τεράστια. Πώς θα τραφεί ο πληθυσμός αυτός, πώς θα διασφαλίσουμε την προστασία τους. Μαθαίνουμε επίσης ότι υπάρχει βία σε βάρος κυρίως των γυναικών στους καταβλισμούς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε, πιστεύετε ότι υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν? 865 εκατομμύρια ευρώ έχετε εξοδέψει από τον προπολογισμό σας για τη Συρία για 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Πώς θα τα βγάλετε πέρα μια που εμείς συνεισφέρουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο όταν οι πρόσφυγες αυτοί θα έχουν γίνει 3,5 εκατομμύρια και όταν συγχρόνως έχουμε και την αποσταθεροποίηση στο Λίβανο που προβλέπετε. Πρέπει να σας πω ότι θαυμάζω πολύ το έργο σας στον ανθρωπιστικό τομέα που είναι τόσο δύσκολος, αλλά δεν μπορώ παρά να σας το ρωτήσω. Ποια είναι η αντίδρασή σας στην ταινία Ασιστός Μορτέλ στην IT που δείχνει οι τοπικές αρχές ότι τελικά δεν συνέβαλαν καθόλου στο έργο αποκατάστευσης και στην ε, βοήθεια. Είναι μια ταινία η οποία πραγματικά σόκαρε τον πληθυσμό. Θέλω τις απαντήσεις σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κόρτες, Κόρτες Λάστρα που υποστηρίζει την χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και των πολιτών μας, στην πρόταση που έχει υποβληθεί έχουμε μικρή αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και όχι μείωση. Αρκεί η μικρή αυτή αύξηση για να ε, αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες. Το μέλλον θα μας δείξει, αλλά τουλάχιστον έχουμε αυξήσει τις πιστώσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια και έχουμε αυξήσει λίγο το αποθεματικό επίγουσας βοήθειας. Εγώ θα ήθελα να έχω δει μεγαλύτερη αύξηση εδώ, ίσως το Κοινοβούλιο να μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον πρέπει να υπερασπιστούμε την ευελιξία όσον αφορά την ακατανομή πόρων στα μέσα που έχουμε για την εξωτερική δράση. Για να σας εξηγήσω πόσο, ε, πόσο μεγάλη σημασία αυτός είναι αυτό. Πέρσι ήταν ε, τρομερή χρονιά. Είχαμε την κρίση στη Συρία, είχαμε την ε, νομισματική κρίση ε, και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου είχαμε σοβαρά προβλήματα. Λόγω της δικής σας υποστήριξης, της υποστήριξης του Κοινοβουλίου και της αρχής του προπολογισμού και της Επιτροπής, μπορέσαμε να αναδιαθέσουμε πάνω από 200 ευρώ από το μέγιστο του προϋπολογισμού μας στο αποθεματικό ε, ε, επίγουσας ανάγκης, το οποίο ανέρχεται σε 1,1 δις, ενώ τελικά ε, καταλήξαμε με 1,3 δις και έτσι καταφέραμε να βρισκόμαστε μπροστά και για τους ανθρώπους ε, στη ζώνη Σαχέλ. Ε, τα εκατομμύρια αυτά ε, έκαναν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Μπορεί να μην το είδαμε στις ειδήσει ως μεγάλη κρίση, αλλά θα μπορούσε να είναι. Εμείς ενεργήσαμε προαιρετικά. Βέβαια, ε, είναι ρόλος μου ως επίτροπος να ε, αγωνίζομαι για τα θέματα αυτά, όπως ε, και για την επιτροπή σας είναι. Εάν λοιπόν μπορείτε να αυξήσετε το αποθεματικό επίγους ανάγκης, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά να αυξήσετε και τη δυνατότητά μας, τη δυνατότητά μας για ανακατανομή των πόρων στο μέλλον, ανάλογα με τις προτεραιότητες. Και χρησιμοποιώ τον όρο ευελιξία. Ευελιξία για μας είναι τεχνικός όρος, αλλά για ένα παιδί που ε, αγωνιά να επιβιώσει ε, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Και ε, δεν δραματοποιώ τα πράγματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας παρακαλώ λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή την ευελιξία και αν κάνετε σκληρή δουλειά όσον αφορά το αποθηματικό, ε, εμείς προτείναμε 350 ε, εκατομμύρια, τα κράτη-μέλη ε, το μείωσαν αυτό σε 280, είπαν ούτως ή άλλως είναι παραπάνω από 250 που είχαμε πριν. Εγώ θα έλεγα όμως ότι τα 350 εκατομμύρια είναι περισσότερα από τα 280 και στο παρελθόν είδαμε ότι το αποθεματικό αυτό είναι ζωτική σημασία για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και ηθικά αλλά και προς το δικό μας συμφέρον. Ε, διότι πρέπει να ε, σκεφτούμε τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε ενεργήσει αποφασιστικά στην περίπτωση του Μαλή. Ε, όχι μόνο για το Μαλή, αλλά ε, και γενικά στη ζώνη Σαχέλ. όσον αφορά την παρατήρηση του κυρίου Γκέρενς για τις ευρωπαϊκές δράσεις στα κράτη-μέλη. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προοδεύσει όσον αφορά τον εξετάζουμε τη γενική εικόνα μαζί με τα κράτη-μέλη. Τη γενική εικόνα όσον αφορά τις κρίσεις. καλέσαμε την ΚΟΧΑΦΑ, την Ομάδα Εργασίας για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει μια επίγουσα κατάσταση, ε, συγκαλούμε ε, συναδρίαση ε, και ζητάμε συντονισμένη δράση. Όσον αφορά τη Συρία, αυτό είναι υψίστης σημασίας Ε, διότι οι συλλογικοί μας πόροι δεν αρκούν και μόνο η αναγνώριση ότι συλλογικά μπορούμε να καταφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεσμευτήκαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ως Κομισιόν και κράτη-μέλη, ε, να διαθέσουμε 370 ε, εκατομμύρια δολάρια μια υπόσχεση που τηρήσαμε. Βλέπουμε όμω ότι υπάρχει και συμπληρωματικότητα όσον αφορά τι δράσει μα. Φροντίζουμε να υπάρχει συμπληρωματικότητα ώστε να μην χρηματοδοτούμε έναν τομέα, να μην υπερχρηματοδοτούμε έναν τομέα και να μην χρηματοδοτούμε άλλου. Ε, η συνεργασία αυτή λοιπόν ε, βελτιώνεται. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, το βλέπουν αυτό. Ο Κλάους ε, που είναι ο Γενικός Διευθυντής θεωρεί ότι αυτά είναι πόρια για όλους. Έχουμε ε, πολλούς ανθρώπους ε, στα ε, στα καυτά σημεία των σαγωγικών του πλανήτη και απομένει πολλής δρόμος ακόμα για μας, αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν και φυσικά θα πρέπει να προσπαθούμε να, βελτιώσουμε να τα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερα όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα με την πολιτική πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όσον αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση, έχουμε ε, κρατήσει πολύ απλή θέση. Λέμε ότι είμαστε μέσα, αλλά είμαστε και έξω. Είμαστε μέσα επειδή φυσικά όλοι ζούμε στον ίδιο πλανήτη. Η πολιτική δράση μπορεί μπορεί να είναι εις βάρος κάποιου. Το τι θα βοηθήσει ή το τι θα βλάψει κάποιον ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητιέται ε, γι' αυτό συνεργαζόμαστε και παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε οποιαδήποτε κρίση. Αλλά οι αποφάσεις ε, για την ανθρωπιστική δράση λαμβάνονται με βάση δύο θέματα, τις ανάγκες και την ε, πρόσβαση στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεν παίζουν εδώ πολιτικά συμφέροντα, είμαστε λοιπόν ανεξάρτητοι και έχετε απόλυτο δίκιο ότι στις επικίνδυνες περιοχές ε, εάν ε, δεν ήμασταν ε, τόσο ανεξάρτητοι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε στη Συρία. Αλλά πάρτε για παράδειγμα τον βορρά του Μαλή. Εκεί Είμαστε παρόντες επειδή είμαστε ουδέτεροι. Τώρα που ε, γίνονται προσπάθειες ανάκτησης του Βορρά. Ποιος είναι παρόν, η ανθρωπιστική κοινότητα. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ έχει διαθέσει 23 εκατομμύρια ευρώ για τους ε, ανθρωπιστικούς οργανισμούς για να ξεκινήσει η αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, εκπαίδευση, ε, ηλεκτρικό και νερό επειδή είμαστε παρόντες. Δεν θα ήμασταν παρόντες όμως εάν ε, είχε θεωρηθεί ότι ε, κρατάμε πολιτική θέση, κάποια πολιτική θέση. Ε, προς όφελος ε, όλων λοιπόν προσπαθούμε να είμαστε ουδέτεροι και ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι. Πώς λειτουργούν λοιπόν όλα αυτά. Ειλικρινά, μερικές φορές ε, βρισκόμαστε στη λάθος θέση. Είμαστε εκεί, ξέρουμε τι χρειάζεται, ε, ε, αγωνιζόμαστε να πετύχουμε, να γίνουν κάποιες δράσεις. Αντί να κουνάει ο σκύλο στην ουρά του, είναι σαν να προσπαθεί η ουρά να κουνήσει το σκύλο και είναι λίγο δύσκολο αυτό. Το πρόβλημα είναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ναι, επειδή είμαστε κοντά στα προβλήματα. Πάρτε τη Συρία για παράδειγμα. Στο Λίβανο, στη Γιορδανία, βλέπουμε πόσο απειλεί τη σταθερότητα του Λίβανου και η Γιορδανία η ροή των μεταναστών. Βλέπουμε πώς οι κοινότητες στρέφονται κατά των Συρίων, οι κοινότητες που, του που τους δέχονται λόγω του μεγάλου αριθμού τους και του ανταγωνισμού ε, για θέσεις εργασίας, ε, για υπηρεσίες υγείας, ε, εκπαίδευση κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε για περισσότερους πόρους, περισσότερη πολιτική δράση για να σταθεροποιήσουμε τη Ιορδανία και το Λίβανο. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στα θέματα αυτά. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι αρνητικό ότι βρισκόμαστε εκεί πριν από όλους. Ε, ως υπηρεσία είμαστε υποχρεωμένοι ε, να το κάνουμε αυτό. Ε, υπάρχει όμως η εφαρμία που λέει ότι μπορεί κανείς να πάει το άλογο ε, στο πηγάρι, δεν μπορεί να το κάνει να πιει όμως. Ε, και εκεί απελπιζόμαστε μερικέ φορέ. έχουμε το άλογο, είναι, δίπλα, είναι μπροστά η πηγή, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Θα ήθελα όμως ε, να τονίσω και όλας ότι όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε σε περιπτώσεις κρίσης, τόσο βελτιώνονται οι δυνατότητες συνεργασίας μας. Ε, το Μάλι είναι εξαιρετικό θετικό παράδειγμα. Συμμετείχαμε ήδη από την αρχή. Συμμετείχαμε στη διαμόρφωση της ε, της ε, δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί οι στρατιώτες λοιπόν ε, πήγαν εκεί για να πολεμήσουν αλλά και για να προστατεύσουν ε, τους πολίτες. Όσο λοιπόν βασιζόμαστε στις επιτυχίες μας, τόσο περισσότερες ελπίδες έχουμε να έχουμε συμπληρωματικότητα, να έχουμε ισχυρό δυναμικό και να εργαζόμαστε προς όφελος όλων. Και αυτό ουσιαστικά με φέρνει στην ελληνική και συνεργασία. στον κόσμο μας ε, δεν ε, είναι οι φτωχές χώρες ε, ευάλωτες και οι πλούσιες χώρες προστατευμένες. Στην Οκλαχώμα είδαμε τους τυφώνες, είδαμε την τριπλή καταστροφή στη Ιαπωνία, είδαμε στο Μανχάταν τον τυφώνα Σάντι, βλέπουμε την αλλαγή του κλίματος. Οι κίνδυνοι αυξάνονται για όλους. Θεωρούμε μέρος της εντολής μας να προετοιμαστούμε, να προλάβουμε, να συνεργαστούμε και με άλλους όμως, να έχουμε γενική αλληλεγγύη. Δεν είναι τελείω απίθανο κάποια μέρα μια πλούσια χώρα να χρειάζεται βοήθεια. Η Ιαπωνία χρειαζόταν, χρειάστηκε βοήθεια, το Μανχάταν χρειάστηκε βοήθεια. Η οικοδόμηση αλληλεγγύη λοιπόν ε, δεν έχει να κάνει μόνο με το δισεκατομμύριο των ανθρώπων που κοιμούνται πεινασμένοι. Έχουμε φτωχέ ευάλωτε χώρε, ε, αλλά χρειαζόμαστε αλληλεγγύη επειδή ε, υπό το φως της αλλαγής του κλίματος, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα είναι ε, να ε, ε, έχουμε αλληλεγγύη, να έχουμε μια κοινή πλατφόρμα δράσης. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Ε, καταλαβαίνω αυτό που είπατε περί προβλέψεων, περί προορατικότητας. Γι' αυτό έχουμε το νέο κέντρο ε, στόχος μας ε, είναι να έχουμε ε, περισσότερο δυναμικό για να προβλέπουμε τις κρίσεις, τις κρίσεις και μακριά από μας, αλλά και κοντά σε μας Και η απάντησή μου προς εσάς είναι συνεχίστε να μας πιέζετε για να δούμε πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε καλύτερα το δυναμικό μας για να μπορούμε να προβλέπουμε καταστροφές και να ενεργούμε συλλογικά. Ε, προσπαθούμε να ε, επικοινωνούμε με χορηγούς. Ε, είχα πάει στα κράτη του κόλπου, στην Κίνα, τη Ρωσία, δεν έχω πάει ακόμα στην Βραζιλία. Αλλά αν ανανεωθεί η θητεία μου θα πάω. Και είναι δύσκολο αυτό διότι... Ε, υπάρχουν διαφορετικές προοπτικές, αλλά αδύνατον δεν είναι, διότι υπάρχει ένα τομέας στην πρόληψη και αντιμετώπιση των κρίσεων, όπου ευτυχώς δεν υπάρχει πολιτική. Είναι ένα ε, θέμα στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτόν τον έναν τομέα για να οικοδομήσουμε πιο αποτελεσματική συνεργασία και να επενέσουμε όσους κάνουν ε, σωστά πράγματα. Το Κουβέιτ ε, οργάνωσε την διάσκεψη για τη Συρία, ε, υποσχέθηκε 300 εκατομμύρια δολάρια ε, και τα παρέδωσε. Τους επενώ όπου και να πάω. Και ενθαρρύνω και άλλους να κάνουν το ίδιο, διότι δεν το κάνανε αυτό όλοι. Ε, καλό λοιπόν και άλλους να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Όσον αφορά τους ε, πρόσφυγες Λόγω της αλλαγής του κλίματο. Ε, έχουμε λοιπόν τώρα μια πολιτική όσον αφορά την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Έπρεπε να την είχαμε πολύ πιο πριν, ε, αλλά τώρα την έχουμε. στον τομέα λοιπόν της ανθρωπιστικής βοήθειας... Προσπαθούμε να πετύχουμε προστασία από κλονισμού ιδιαίτερα όσον αφορά το κλίμα, ε, με τη χρηματοδότησή μας. Ε, ο Επίτροπος Πίμπαλξ και εμείς ο Επίτροπος Πίμπαλξ ως ε, μεγαλομέτοχος και εμείς ως πιο μικροί μέτοχοι έχουμε χρηματοδοτήσει δύο πολύ μεγάλα προγράμματα, 1,5 δις για την προετοιμασία στη ζώνη Σαχέλ ε, και στο κέρας της Αφρικής. με στόχο να, να πανίσουμε συνολικά ένα τίστα μέσα στην επόμενη επταετία. Παίρνουμε λοιπόν, ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα η αλλαγή του κλίματος ε, και η προσαρμογή σε αυτό. το θέμα αυτό οδηγεί σε εκτόπιση περισσότερων ανθρώπων, σε πρόσφυγες. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να βοηθήσουμε κοινότητες με απλά μέτρα, ώστε να μπορούν να αντέξουν ε, ε, σε, ε, στους κίνδυνους που προκαλεί η αλλαγή του κλίματος ε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε αρκετά μεγάλη κλίμακα δεδομένη ε, τη ε, τεράστια κλίμακα του προβλήματο. Όσον αφορά τη Συρία, κύριε Ζολή. Είναι τρομερό, ιδιαίτερα για τα παιδιά και ιδιαίτερα για, για τα κορίτσια. Ποιος υποφέρει περισσότερο σε μια τέτοια κρίση. Το 55% των προσφύγων είναι παιδιά κάτω των 18 ετών. και μεταξύ των παιδιών ε, υποφέρουν περισσότερα τα κορίτσια, διότι είναι πιο πιθανό να μην πάνε σχολείο, αν και βλέπουμε και αγόρια που δεν πηγαίνουν σχολείο. Το 20 με 30% των παιδιών ε, σε σχολική ηλικία πηγαίνουν στο σχολείο. Ε, ε, ήταν χώρα μέσου εισοδήματος, ε, είχαν πολύ ψηλό επίπεδο στην εκπαίδευση. Βλέπουμε λοιπόν παιδιά από τη Συρία που δεν πηγαίνουν σχολείο, μια χαμένη γενιά. Και κάθε φορά που ταξιδεύω, πάντα βλέπω αυτά τα πρόσωπα τα οποία δεν μου φεύγουν από το μυαλό. Να σας πω μια ιστορία από το τελευταίο μου ταξίδι. 13 χρονών είναι η Άισα, η μητέρα της ε, είναι ανάπηρη, η Άισα δεν πηγαίνει σχολείο, διότι είναι η μόνη που μπορεί να εργαστεί και να βγάλει χρήματα στην οικογένεια. Εργάζεται λοιπόν και βγάζει λιγότερο από 2 ευρώ την ημέρα. Εργάζεται στα χωράφια. Μιλώ λοιπόν με την Άισα και τη μητέρα της και ήθελα να πω ότι ελπίζω ότι θα ξαναγυρίσει στο σχολείο και ήξερα ότι δεν θα επιστρέψει. Δεν μπορούσα να της ε, πω ψέματα. Ξέρω τι θα γίνει. Θα παντρευτεί νωρίς, θα παντρευτεί μάλλον στα 14 και εκεί θα τελειώσουν τα όνειρά της. Υπάρχουν χιλιάδες κορίτσια σαν κι αυτήν. Τα κορίτσια παντρεύονται νωρί διότι τελικά ε, εκείνα αποτελούν ε, πηγή εισοδήματος για τις απελπισμένες οικογένειές τους. Και πολιτιστικά είναι πιο εύκολο αποδεχτό αυτό εκεί από ότι είναι για μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα της ζωής. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, ε, να δώσουμε προτεραιότητα στο Λίβανο και στη Ιορδανία, βοήθεια προς τις ε, τοπικές κοινωνίες, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ε, απορροφούν πρόσφυγες, να διαβρύνουν τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας. Τρία εκατομμύρια πρόσφυγες δεν είναι καθόλου αδύνατο να δούμε. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε να έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση, όχι όμως ε, μόνο από ανθρωπιστικές πηγές, ε, αλλά και από ε, πηγές αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό που με απογοήτευσε περισσότερο στο Λίβανο Ε, ήταν η Παγκόσμια Τράπεζα. Η... Παλιά δούλευε για την Παγκόσμια Τράπεζα. Αλλά πού ήταν, ήταν απούσα, παρότι ε, ο Λίβανος ε, αποτελεί προτεραιότητα όσον αφορά τις χώρες που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να μην επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στην πολιτική λύση που θα δοθεί εντό τη Συρίας, διότι ακόμα και αν έχουμε μια τέτοια λύση αύριο, ήδη η κρίση αυτή έχει κρατήσει πολύ και γι' αυτό Πρέπει να υποστηρίξουμε το Λίβανο και τη Γιορδανία και να δώσουμε προτεραιότητα στις χώρες αυτές. Όσον αφορά την ταινία για την IT, δεν την έχω δει, πρέπει να το ομολογήσω. Ε, ε, οι συνάδελφοί μου την έχουν δει, εγώ δεν την είδα, οπότε δεν μπορώ να σας εκφράσω γνώμη. Αλλά μπορώ να σας πω ότι είδα στην IT πριν ε, τρία χρόνια και τώρα τρία χρόνια μετά. Όσο τρομερή, όσο τρομερός και να ήταν ο σεισμός, δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της IT. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου ε, κυβερνητικό δυναμικό. Ο λαός ε, είναι πολύ δυνατός, ε, πολύ αθεκτικός, οι κοινότητες βοηθούν η μία την άλλη, οι αρχές όμως είναι πάρα πολλοί ασθενεί και η έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντι στην κυβέρνηση είναι η μεγαλύτερη που έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Κυρία Ζολή, πριν τρία χρόνια και τώρα, ο κόσμος μου λέει μη δίνετε λεφτά στην κυβέρνηση. Τόση έλλειψη εμπιστοσύνη. τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση κυβερνητικού δυναμικού. Δεν ξέρω τι δείχνει η ταινία. Εγώ όμως, αμέσως μετά το σεισμό, δώσαμε 10 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ. Τρία χρόνια μετά 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ε, συγγνώμη. Εμείς θέλαμε ε, να έχει οικοδομηθεί η χώρα τρία χρόνια μετά. Πώς μπορεί να απορροφήσει κανείς 10 ε, δισεκατομμύρια ευρώ από μια χώρα διαφθαρμένη υπό τον Papa Doc και τον Baby Doc. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη ρεαλισμού όσον αφορά την προσέγγιση μας στην Αιτή. και υπάρχει μεγάλος βαθμός υποκατάστασης ε, της ε, τοπικής διακυβέρνησης ε, από την καλή βούληση των ανθρώπων. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μεταμορφώσει τη χώρα. 10-15 χρόνια οικοδόμησης θεσμών θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τη χώρα. Εγώ φοβόμουν ότι θα ξεχάσουμε την IT επειδή ξεχνάμε γρήγορα και αυτό θα ήταν τεράστιο λάθος θα δω την ταινία και ε, υπόσχομαι να σας πω την πραγματική μου γνώμη αντί να σας διαβάσω τις σημειώσεις που μου δώσαν οι συνεργάτες μου. Ευχαριστούμε. Η κύριε Στίχλερ Ναι, απάντησε στην ε, ερώτηση. Καλώς, λέει η κυρία Ζολή, πρόεδρος. Έτσι τελειώνει η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στα πλαίσια αυτού του διαφρομένου διαλόγου. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιώργεβα που ήταν εδώ μαζί μας και που συμμερίστηκε μαζί μας τις απόψεις της όπως κάνει πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Oh, wait. Yeah. You're going to answer me? Yes. Yes. Okay. But you already answered it. Okay. This lack of competence, I think. Yes.